Uh, Καλημέρα σας. Ξεκινάει η ψηφοφορία και θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσουμε ε, την, ε, τις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία είναι σχετικά με την, ε, το Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού. Λοιπόν, μετά θα έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανή Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μακροχρηματοδοτήσεων για Απασχόληση μετά το κοινοτικό πρόγραμμα Progress ε, και μετά το ε, χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για πέντε λεπτά να περιμένουμε για να έχουμε ε, ε, ε, απαρτία διότι πολλοί συνάδελφοι έχουν καθυστερήσει. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να δώσετε μία περίοδο ο χάριτος πέντε λεπτών παρόλη την ακρίβεια της Προεδρίας ε, κύριε, ε, ήθελα να αρχίσουμε ε, εγκαίρως αλλά εντάξει θα περιμένω μερικά λεπτά και θα δούμε ποιος άλλος θα έρθει ακόμη. Okay, you are ready.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 Έχετε τις κάρτες σας γιατί θα πρέπει χωριστά να μετρήσουμε όσους δεν έχουν κάρτα. Έχετε όλη την κάρτα σας. Λοιπόν, προχωράμε στην ε, πρώτη ψηφοφορία, η οποία είναι αριθμός 18.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 Uh, uh, λοιπόν, 17 uh, υπέρ, καμνής κατά και καμία αποχή. Σας παρακαλώ, καθίστε διότι ψηφίζουμε εφόσον λοιπόν υπήρχε συντριπτική πλειοψηφία θα προχωρήσουμε εις ε, την ψηφοφορία διανατήσεως χειρός. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Είσαστε όλοι υπέρ. Ε, κατά. Εγκρίνεται καταπίπτει 41, η 42, στη 43 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται καταπίπτει η 19, η 44, 45. Ψηφίζουμε την 20 από την εισηγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 καταπίπτει 23 αποσύρεται 47 υπέρ κατά καταπίπτει η 24 αποσύρεται η 48 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 48. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ψήφισαν 42, 16 υπέρ, 26 κατά, καμία αποχή, ε, απορρίπτεται. 25 και 26 θα ψηφιστούν αργότερα γιατί ε, θα, ε, ε, θα καταπέσουν αν η πρώτη συμβιβαστική αποτύχει. 20 η ένα της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ Κατά. Θα χρειαστεί να ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία σχετικά με τη συμβαστική υπαριθμών 1. Λίγοι. ψήφισαν 42, 26 υπέρ, 16 κατά, 27 μάλλον υπέρ και 16 κατά. Με συγχωρείτε κύριε Σρότερ, αλλά δεν σας είχα μετρήσει. 25 και 26 καταπίπτουν και πάμε στην, ε, στην 27 γιατί καταπίπτει και η τροπολογία 2 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 καταπίπτει Μάλλον όχι. Ε, θα ψηφιστεί αργότερα εάν υιοθετηθεί η συμβαστική 2 ή 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά Ας κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Ξεκινάει η ψηφοφορία σχετικά με την 29. Ε, Λίγη. ψήφισαν 43, 19 υπέρ και 24 κατά. 4 που συνάδει με την 30 υπέρ κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει. Λίγοι. Ψήφισαν 43, 18 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αντικαθιστά την 6 και την 31 που καταπίπτουν 7 της συγγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 της συγγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33, 9 και 34 καταπίπτουν, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά. Για να ξαναδούμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. οι 10 και οι 28 καταπίπτουν, συμβιβαστική 5 που αντικαθιστά την 35 και την 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρα καταπίπτουν 35 και η 11 συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, καταπίπτει 12 και η 36 και υπάρχει μία ε, φορική τροπολογία της εισηγήτριας υπαριθμών 37. Υπάρχει καμία αντίθεση, ε, <clears throat> το έχετε στα χαρτιά σας. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38, πάλι ψήφο τροπολογία προφορική της ε, εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ας ελέγξουμε ξεκινά ε, η ψηφοφορία για την τροπολογία 38 ε, με την προφορική τροπολογία Λίγη. Ψήφισαν 46, 26 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Και προχωράμε τώρα στην 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται οι 14 και 39 καταπέφτουν, 15 της ηγήτρες υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά. Αποχές Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάμε για την τροπολογία 40. Κλείνει. Ψήφισαν 45. 28 υπέρ, 14, 15 κατά, εγκρίνεται. Η 17 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ξεκινάει. Λίγη ψήφισαν 45, 46, 45 υπέρ και μία αποχή. Ε, και συγχαίρω τη Μάριαν Χάλκιν. Με μία ψηφοφορία μόνο. Ποιος είναι υπέρ. 20-10 κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Uh, Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα χθε. Γιατί στι 9.30 θα αρχίσει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών. Και ακόμη δεν είμαστε βέβαιοι ότι ολοκλήρωσαν την ψηφοφορία. Γι' αυτό συζητούμε περί τη ακολουθητέα διαδικασία. Αλλά παρακαλώ παραμείνετε στην αίθουσα γιατί εντό ολίγου θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Απλώ προσπαθούμε να μάθουμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών που δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Uh, Έχω μία πρόταση να σας υποβάλω. Θέλω τη συμβουλή σας ως προς την πρόταση που θα σας κάνω. Εγώ θα έλεγα να περάσουμε στην ψηφοφορία, να συνεχίσουμε. Υπάρχει μια ενδεικτική να κάνουμε μια ενδεικτική ψηφοφορία για τι ε, τροπολογίε τη Επιτροπή Προπολογισμών. Αν καταψηφιστούν στην Επιτροπή Προπολογισμών, φυσικά δεν πρόκειται να τι ψηφίσουμε εμεί. Θα είναι ενδεικτική η ψηφοφορία μα για τι τροπολογίε τη Επιτροπή Προπολογισμών. Η σημαντική ψηφοφορία είναι η δεύτερη για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Progress για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Έχουμε πολλές τροπολογίες για το πρώτο θέμα. Οπότε μέχρι να φτάσουμε στο πρόκρες θα έχει αποσαφινιστεί η κατάσταση. Συμφωνείτε να έχουμε ενδεικτική ψηφοφορία για τις τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών, περιμένοντας την έκβαση στην ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ας ε, αρχίσουμε την πρώτη μας ψηφοφορία. Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων Progress. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Οικονομικών. Ε, τροπολογία 5. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία εκών υπαριθμών 5. Τέλος ψηφοφορίας. 46, 18 υπέρ, 27 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται η τροπολογία 5. Πρώτη τροπολογία Επιτροπής Προπολογισμών. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 49 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 49 παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 46, 18 υπέρ, 28 κατά και καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 8, 51, 52 και 53 καταπίπτουν. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 έχει αποσυρθεί. Η 55 καταπίπτει εφόσον έχει εγκριθεί τροπολογία 1. Το ίδιο 56, 57 αποσύρεται, 58, 59 καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν οι 10, 60, 61, 62, 63, 64 και 65. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 66 έχει αποσυρθεί. 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ενδεικτική ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ για την τροπολογία 5 της Επιτροπής Προπολογισμών. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 68 έχει αποσυρθεί. 69. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 70 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 71 Τέλος ψηφοφορίας. 46 ψήφισαν, 20 υπέρ, 25 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 72. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 46 ψήφισαν, 13 υπέρ, 33 κατά, χωρίς αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 75, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 14, 77, 78 ψηφίζουμε. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 46, 26 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 45, 7 υπέρ, 38 κατά. Καμία εποχή. Δεν είδα πώς ήταν κατά, νόμιζα ότι χρειαζόταν έλεγχος. 12 τροπολογία της Επιτροπής Οικονομικών. Δεν είναι ενδεικτική. Τροπολογία 12 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Λέξη. Ψήφισαν 47, 20 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, επαναλαμβάνω, για την τροπολογία 15 ηλεκτρονικά. Ελπίζουμε ότι άρχισε τουλάχιστον η ψηφοφορία. Τέλος. 45 ψήφισαν, 26 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 82. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 47 ψήφισαν, 26 υπέρ και 20 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αν δεν κάνω λάθος. 84. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 90 άρχεται η ψηφοφορία τέλος Ψήφισαν 47, 24 υπέρ και 23 κατά. Εγκρίνεται. 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 44 ψήφισαν, 26 υπέρ και 18 κατά. Εγκρίνεται. 13. Τροπολογία της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αποσύρεται η 18. η 92, 93, 94 και 95 καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 19 έχει αποσυρθεί. Η 99, 96, 97, 98, 100 καταπίπτουν. Η 20 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 102. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 47 ψήφισαν, 26 υπέρ και 21 κατά. Εγκρίνεται. Η 101 έχει αποσύρθει. 15 τροπολογία της ΕΚΟΝ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κα... Απορρίπτεται. 103. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 τροπολογία Ποιο είναι υπέρ για το θεωρώντας κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Προφορική τροπολογία της κυρίας ε, εισηγήτριας. Υπάρχουν αντιρρήσεις μήπως? Όχι. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία για το αιτιολογική σκέψη αναλφανέ. Ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία 6 άρχεται η ψηφοφορία τέλος 46 ψήφισαν, 41 υπέρ και 5 κατά. Εγκρίνεται. 22, οι 2, 22, 23, 23 24, 25 καταπίπτουν. 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 46 ψήφισαν, 18 υπέρ, 24 κατά και 4 αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 έχει αποσυρθεί. 27, 28, 29 και 30 καταπίπτουν. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4, 31, 32, 33 και 88 καταπίπτουν. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 37 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψήφισαν 45 16 υπέρ 28 κατά και μία αποχή απορρίπτεται Τροπολογία 38. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Οι 1476 καταπίπτουν. Τροπολογία 39. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 10. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 5, 41, 42, 44, 45 και 46 καταπίπτουν. 43. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 6, 47 και 48 καταπίπτουν. Δεύτερη τροπολογία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αναδεικτική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, οχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης, όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 46, 41 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι μάλλον ηλεκτρονικά και αυτή η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 47 ψήφισαν, 42 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται και το νομοθετικό ψήφισμα. Συγχαρητήρια κυρία Ισηγητρία. Θα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα για να δούμε πώς ψήφισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών για να πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Σας παρακαλώ μην απομακρυνθείτε γιατί μπορεί να πάρει μόνο λίγα λεπτά. Μη σας πω και λίγα δευτερόλεπτα. Μιλάμε στο τηλέφωνο με τον τελικό λογισμό.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 Uh, ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά θα λάβουμε γρήγορα την, αποφασή μας. Αν δεν έχει ψηφίσει η Επιτροπή Προπολογισμών, νομίζω ότι καλό θα είναι να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε ως ενδεικτική ψηφοφορία και πάλι. Αλλά να περιμένουμε κανένα δύο λεπτά ακόμα για να δούμε μήπως έχουμε νέα από την Επιτροπή προπολογισμών. Ιδάλω λέω να ψηφίσουμε ενδεικτικά, όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Από ό,τι κατάλαβα γίνεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν θα πάρει πολλή ώρα. Περιμένουμε και την τελική επιβεβαίωση. Ψήφισαν πάντως και θα μάθουμε τα αποτελέσματα σύντομα.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

Ακόμα περιμένουμε γιατί θα πρέπει να δούμε αν ψηφίστηκαν οι τροπολογίες από την Επιτροπή Προπολογισμού. I do apologize for this, uh, but we are still waiting. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά περιμένουμε ακόμα. Και επειδή είχε ήδη ψηφίσει η ολοκληρώση τη ψηφοφορία η Επιτροπή Προπολογισμών, νόμιζα ότι ε, καλό αυτό να περιμένουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε κι άλλο. Τι θα κάνουμε, λοιπόν. Αν σε κανένα δύο λεπτά δεν έχουμε νέα, θα ψηφίσουμε ενδεικτικά. Φυσικά, αν έχουν καταψηφιστεί οι τροπολογίες της Επιτροπής Προπολογισμού, δεν θα έχει σημασία το τι θα ψηφίσουμε εμείς εδώ. Αν δεν λάβουμε μία απάντηση σύντομα, θα προχωρήσουμε σε ενδεικτική ψηφοφορία, αν συμφωνείτε. There is somebody running towards... Βλέπω να μας πλησιάζει κάποιος τρέχοντας την ώρα που σας μιλάω.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 Λοιπόν, από την Επιτροπή Προπολογισμών τα νέα είναι τα εξή. Δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία. Στις 11 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία η τροπολογία υπερθμών 3 της Επιτροπής Προπολογισμών έχει τροποποιηθεί, άρα δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Θα προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει εμείς, να μην ψηφίσουμε όμως καθόλου τις τροπολογίες της Επιτροπής Προπολογισμών. Συμφωνείτε? Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνείτε? Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε αλλάζουν τα πράγματα την ώρα που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τροπολογία υπεριθμών 3. Υπέρ. Η τροπολογία 3 παρακαλώ υπέρ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο έλικα, δεν κάνω λάθος. Mrs. Moran, are you ready? Είστε έτοιμη κυρία Μαράν. Uh, Mr. Organo. Κύριε Σοργκάνο, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ανακοινώσω απλά ότι η τροπολογία υπαριθμών 3 έχει αποσυρθεί. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ. Αποσύρθηκε λοιπόν η παριθμόν 3. Τη 3 του προϋπολογισμού δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 1 στο εκτιμώντας 3. Παραμένει ή έχει αποσυρθεί και αυτή. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Θέλετε το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από την τροπολογία αυτή. Θα ήθελα να αποσύρω το όνομά μου από την ε, τροπολογία 2. Αυτά στα συνθήκα θα ζητούσα από το ΕΛΚ να απόσχει από την ε, τροπολογία. Ωραία, να ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τη τροπολογία 1 τη Επιτροπή Προπολογισμών δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε, ούτε την 2 τη επιτροπή Προπολογισμών. Δεν πέρασαν τροπολογίε να ψηφίσουμε το σχέδιο νομοθετική πρόταση πρότασης, νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Everyone voted. Ψηφίσατε όλοι. Αν ψηφίσατε όλοι, τη ψηφοφορία. 45 ψηφίσατε 41 ε, ψηφί υπέρ, 4 κατά, εγκρίνεται συγχαρητήρια. Uh, now we have uh, the motion for resolution. Τώρα έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος, μία ψήφος. Έναρξη ψηφοφορίας. Έναρξη ψηφοφορίας για το σχέδιο ψηφίσματος. Έναρξη ψηφοφορίας, επαναλαμβάνει η Πρόεδρος, για το σχέδιο ψηφίσματος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 44 ψήφοι, 42 υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Πέρασε. Λοιπόν, εγκρίνεται. Uh, that the votes. Και έτσι ολοκληρώνουμε τις ψηφοφορίες μας για σήμερα. Συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στις ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Κυρία Γκάντς, ίσως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Θα πρέπει να συζητήσουμε την ε, εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος ε, τρόπος για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Θα σας πω λοιπόν τι σκοπεύουμε να κάνουμε στις διαπραγματεύσεις, κατά πόσο θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση κτλ. Η Σουηδική Προεδρία φυσικά θέλει να γίνει συμφωνία, να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αλλά να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας πει και την άποψή της. Αν συμφωνείτε δηλαδή με, το, με τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και λυπάμαι που προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το τι θα γίνει στην ψηφοφορία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και καθόμαστε και συζητάμε, αλλά τι να γίνει. Εντάξει, νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Σουητική Προεδρία. Έχουμε ήδη κάνει μία συνάντηση και θα επακολουθήσουν και άλλες. Θα γίνουν και κάποιες ανεπίσημες συναντήσεις και είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τους πόρους και επί του περιεχομένου. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος να αποφασίσουμε για τη σύνθεση τώρα της ομάδας των διαπραγματευτών. Έχουμε μία πρόταση εδώ μπροστά. Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης είναι ο, η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, η συγγήτρια. Και από τις βασικές ομάδες έχουμε δύο προβλήματα όμως, ότι το, το EFD και οι μη εγγεγραμμένοι δεν έχουν δηλώσει Ποιο θέλει να τους εκπροσωπήσει, ποιο θέλει να τους εκπροσωπήσει στις διαπραγματεύσεις. Ίσως θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν λοιπόν. Είστε όλοι υπέρ τη ομάδα αυτή των διαπραγματευτών. Όλοι ξέρετε ποιον έχετε προτείνει για την ομάδα. Έχετε κάποιο πρόβλημα λοιπόν με τη σύνθεση τη ομάδας. Όχι. Σύμφωνείτε όλοι. Εντάξει. Να εξετάσουμε τώρα την εντολή της ομάδας διαπραγμάτευσης. Θα ανακοινωθεί ο τριμερής διάλογος και η γραμματεία του Συμβουλίου θα παράγει ένα κοινό έγγραφο για τις ε, θέσεις των ε, άλλων θεσμικών οργάνων. Το Συμβούλιο ε, προγραμματίζει δύο συναντήσεις. Νομίζω ότι η κυρία Γκόνς είναι ενήμερη για την ημερομηνία των δύο συναντήσεων αυτών και ελπίζω να το γνωρίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 16 Νοεμβρίου 7 ε, το απόγευμα και 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Συμφωνείτε όλοι. Και η τελική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτά μέσω επίσημη επιστολής από το Συμβούλιο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για το θέμα αυτό και πάλι σας συγχαίρω. We Και τώρα να περάσουμε στην παρουσίαση της μελέτης «Δείκτες ποιότητος της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». And I give the floor to Mr. Rafael Munoz, να δώσω τον λόγο στον κύριο Ραφάλ του Μόντο στο Επιστήγιο. Και λυπάμαι για την προφορά μου. ναι, όχι, εγώ ζητάω συγγνώμη για τη δική μου προφορά. Θα μιλήσω ισπανικά, αν μου επιτρέπετε. Muchas ε, Σας ευχαριστώ. Έχω 10 λεπτά ή ένα τέταρτο για να μιλήσω, γιατί δεν ε, μου ανακοίνωσε κανεί το χρόνο αγόρευση. 10 με 15 το πολύ, ένα τέταρτο το πολύ έχετε στη διάθεσή σα. Ε, είμαι συνηθισμένο σε πιο μακροσκελεί παρουσιάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα επικεντρωθώ στο βασικό σχεδιάγραμμα της μελέτης και θα προσπαθήσω να αυπνίσω το ενδιαφέρον σα προκειμένου να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη. Αυτό που επιχειρήσαμε στη μελέτη είναι να αναλύσουμε το κατά πόσο έχει νόημα να φτιάξουμε έναν δίκτυ ποιότητας απασχόλησης. Αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο και αν οι υπάρχοντες δείκτες στη βιβλιογραφία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε να αντικατοπτρίζουν ε, σωστά την έννοια της καλής εργασίας ή της ποιοτικής απασχόλησης, που είναι μια πολυδιάστατη έννοια, με πολλές αποχρώσεις. Και σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο αξιολογούμε περίπου 20 δείκτες που έχουμε στη διάθεσή μας και αφορούν την ποιότητα της απασχόλησης. Θα καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα και για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου δείκτη, αλλά και για τη βιωσιμότητα αυτής της κατασκευής, της δημιουργίας του νέου δίκτυ. Έχει νόημα ένας τέτοιος δίκτυς ποιότητας απασχόλησης. Έχει ενδιαφέρον. Η απάντησή μας είναι καταφατική για πολλούς και διάφορους λόγους. Και τους βλέπετε στη διαφάνεια. Ένα σημαντικό τμήμα της ζωής του ο άνθρωπος την περνάει στην εργασία. Γύρω στις 40 ώρες τη βδομάδα περνάει κάποιος που έχει πλήρη απασχόληση. Ένα μεγάλο τμήμα της ζωής του, το 1 τέταρτο του χρήσιμου εβδομαδιαίου χρόνου του τον περνάει στην εργασία. Η οικονομική θεωρία όταν ασχολείται με θέματα ποιότητας εργασίας και ακολουθώντας μια παλιά παράδοση της κλασικής οικονομίας του Άνταμ Σμιθ θεωρεί ότι αρκεί να ληφθεί υπόψη ο μισθός ε, για να χαρακτηριστεί μια εργασία ως ποιοτική. Ή υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη. Αυτό λέει η θεωρία του... των διαφορών των αντισταθμιστικών. Όταν, υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι κακοί όροι, μερικές φορές υπάρχουν υψηλότεροι μισθοί. Αλλά όταν γίνεται αυτή η αντιστάθμιση στην αγορά, διαπιστώνουμε ότι η αντιστάθμιση περιορίζεται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις. Και οι συνδυασμοί είναι πολλαπλή. Έχουμε εργασίες με καλές γενικές προϋποθέσεις και καλούς μισθούς, με κακές προϋποθέσεις και κακούς μισθούς. Συνδυασμό καλών προϋποθέσεων και κακών μισθών ή καλών μισθών και κακών προϋποθέσεων είναι πολύ σύνθετη η κατάσταση. Επίσης, έχουμε την παγκοσμιοποίηση, τον νέο καπιταλισμό και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Με όλα αυτά τα νέα στοιχεία εξετάζεται το κατά πόσο με τις νέες τάσεις η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δημιουργεί αύξηση των θέσεων εργασίας κακής ποιότητας. Έχουμε σαφείς πληροφορίες για το ποιες θέσεις απασχόλησης παραμένουν ή ποιες χάνονται. Δεν υπάρχει κατάλληλος δείκτης για να καταμετρήσουμε αυτή την έννοια της ποιότητας της απασχόλησης. Αν έχουμε ένα τέτοιο ειδικό δίκτυο ποιότητα, θα μπορέσουμε με πιο γενικό και ευρύ τρόπο να αξιολογήσουμε κάποια καθεστώτα απασχόλησης και τις διάφορες αγοράς εργασίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδυάζουν ποιότητα, μισθούς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε διαφορετικά ποσοστά και αναλογίες. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι, όπως σας είπα, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει νόημα να φτιάξουμε έναν ειδικό δίκτυ ποιότητας για να καταμετρήσουμε την ποιότητα της απασχόλησης. Απαντήσαμε λοιπόν στο ερώτημα αν έχει νόημα, αν αξίζει προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου δίκτυ από άποψη κοινωνικής ανάλυσης. Αλλά το θέμα είναι πώς θα κατασκευαστεί ένας τέτοιος δείκτης, πώς θα διαμορφωθεί, ποιες θα είναι οι προσεγγίσεις που θα υιοθετήσουμε. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχολές. Η πρώτη σχολή προσπαθεί να ακολουθήσει ένα σύντομο μονοπάτι, γιατί η έννοια της απασχόλησης είναι προσωπική, δύσκολο να καταμετρηθεί, πολυδιάστατη και πολλές φορές είναι θέμα προσωπικής υποκειμενικής αντίληψης του εργαζόμενου για το πώς αντιλαμβάνεται την εργασία του. Εδώ βλέπετε στο γράφημα ένα δίκτυο ικανοποίηση ε, με την εργασία πολλών χωρών με βάση μία έρευνα του 2005. Απλώς ρωτώ με τον εργαζόμενο αν είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά του. Εδώ βλέπουμε στα αποτελέσματα ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίηση ε, με τη εργασία και μια μικρή διακύμαση στην ικανοποίηση μεταξύ των χωρών που γνωρίζουμε από άλλε συμπληρωματικέ πληροφορίες και πηγέ ότι έχουν πολύ διαφορετικέ συνθήκε εργασία. Είναι πολλά και διάφορα λοιπόν τα στοιχεία ε, που συνυπολογίζονται. Γι' αυτό είναι δύσκολο να συνδυάσουμε την ικανοποίηση με την εργασία με κάποιους αντικειμενικούς όρους για την ποιότητα της εργασίας. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να μην ρωτήσουμε τους εργαζόμενους αν είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, αλλά να τους ρωτήσουμε ποιους παράγοντες θεωρούν σημαντικούς κατά την αξιολόγηση μιας εργασίας. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό, η ασφάλεια της εργασίας, το εισόδημα, δυνατότητες προαγωγής, αυτονομία, ελαστικότητα του ωραρίου εργασίας. Εκεί βλέπετε στοιχεία από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένε Πολιτείε και 17 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν υπόψη πολλές συνθήκες και όχι μόνο το μισθό ή την ασφάλεια για να αξιολογήσουν τη δουλειά τους και να την κρίνουν καλή ή κακή. Και αυτή είναι μια προοπτική για τη δημιουργία δεκτών ποιότητας. Να επικεντρωθούμε δηλαδή στα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη ο εργαζόμενος για να χαρακτηρίσει τη δουλειά του ως καλή ή κακή. Αλλά υπάρχει και άλλος δρόμος. Να αναλύσουμε την βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών και να δούμε τι μας λένε οι εμπειρογνώμονες τι μας λένε οι κοινωνιολόγοι που ασχολούνται με την απασχόληση. Ποια στοιχεία είναι σημαντικά για την ποιότητα της απασχόλησης, αλλά και έμεσα ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευημερία του εργαζόμενου. Και από τη βιβλιογραφία για τη δουλειά, για την συνεργασία, βλέπουμε ότι εκτός από τους μισθούς λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως η συμμετοχή στον χώρο της εργασίας, η βιομηχανική δημοκρατία, η σημασία που έχουν το στοιχείο, το στοιχείο, το της εξουσίας, ε, της, ε, του νοήματος που έχει δουλειά, η αυτονομία που έχει ο στη δουλειά του, η σταθερότητα της απασχόλησής του. Από τη βιβλιογραφία λοιπόν των κοινωνικών επιστημών μπορούμε να συντάξουμε ένα ολόκληρο κατάλογο παραγόντων που είναι σημαντική για την ε, διαμόρφωση ενός μοντέλου ποιοτικής εργασίας. Και αυτό κάνουμε σε ένα από τα κεφάλαια της μελέτης. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις προοπτικέ, ιδιαίτερα τη δεύτερη προοπτική, να ρωτήσουμε δηλαδή του εργαζόμενους και την τρίτη προοπτική να ρωτήσουμε τους εμπειρογνώμονε και τους κοινωνιολόγους, καταλήγουμε σε ένα γενικό μοντέλο ποιότητα εργασία που στηρίζεται σε δύο άξονες, δύο διαστάσεις, ε, τη διάσταση της ποιότητας εργασίας, ε, work quality, και της ποιότητας απασχόλησης, employment quality που συνοψίζουν ε, πολύ εύστοχα όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία. Και έτσι δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, δίκτυ ποιότητας, αλλά χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο για να αξιολογήσουμε τα υπάρχοντα μοντέλα και τα υπάρχοντα στην αγορά εργασίας. Και σε ό,τι αφορά το work quality, την ποιότητα εργασίας, Βλέπουμε την αυτονομία στην εργασία, τις φυσικέ φυσικές συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται, κάποιες μεταβλητές υγείας, κίνδυνος ατυχήματος, ταχύτητα, το κοινωνικό μέσο στον οποίο διαδραματίζεται η εργασία. Όλες αυτές οι μεταβλητές μπορούν να καταλήξουν σε αντικειμενικούς στόχους για την καταμέτρηση αυτών των στοιχείων που προέρχονται από υπάρχουσες πηγές. Και έχουμε και την employment quality, το, την ποιότητα της απασχόλησης με το είδος της σύμβασης, ε, τις α, ε, ώρες εργασίας, το, το μισθό, τα κοινωνικά επιδόματα, την ελαστικότητα του ωραρίου εργασίας και οι παράγοντες και από αυτές τις δύο κατηγορίες επηρεάζουν την ποιότητα. Έχουμε και κάποια παραδείγματα στην έκθεσή μας. Και έτσι αξιολογούμε το σύνολο των δικτών που υπάρχουν στην αγορά. Πρώτα απ' όλα όμως για να φτιάξουμε ένα νέο δίκτυ θα πρέπει να απαντήσουμε σε μια σειρά θεωρητικών και μεθοδολογικών ε, ζητημάτων. Δεν πρόκειται να τα αναλύσω εδώ. Για παράδειγμα, θα καταμετρήσουμε διαδικασίες ή αποτελέσματα. Η σημασία, σημασία έχει η συμμετοχή ως προς τη διαδικασία ή η συμμετοχή ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τους όρους εργασίας. Θα έχουμε στατικούς δείκτες, όπως είναι τα σημερινά χαρακτηριστικά της εργασίας ή δυναμικ, δυναμικούς δυνατότητες ε, βελτίωσης. Τα στοιχεία θα είναι ατομικά ή ομαδικά ώστε να δούμε αν τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία των χαρακτηριστικών των θέσεων εργασίας συσσωρεύονται σε ορισμένους εργαζόμενους ή κατανέμονται σε πολλούς. Το ίδιο μοντέλο χρησιμεύει για, κάθε, για όλες τις χώρες ή θα πρέπει να εκπονήσουμε διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα σύνθετο δίκτυ ή μια συστοιχεία δικτών 15, 16, 20 δικτών και όχι ένα σύνθετο συνολικό δίκτυ. Αν έχουμε συνολικό δίκτυ, πώς θα γίνει η πρόσθεση, με τι μεταβλητές, όλα αυτά τα μεθοδολογικά και τεχνικά ζητήματα θα πρέπει να τα απαντήσουμε πριν ε, δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυ. ο δείκτης της ποιότητας εργασίας είναι πολυδιάστατος, γι' αυτό και είναι πολύ περίπλοκος. Αλλά ούτως ή άλλως, όταν έχουμε ένα δείκτη, είτε το αντιμάριθμο, είτε του ΑΕΠ, θα πρέπει προηγουμένως έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά τα μεθοδολογικά ερωτήματα. Με αυτό το, αυτή τη θεωρητική ανάλυση και με αυτό το γενικό μοντέλο αναλύσαμε 18 ειδικού ε, δείκτες που έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες, διαφορετικές πόρους, διαφορετική θεσμική στήριξη. Μερικές, μερικοί δείκτες είναι προτάσεις συγκεκριμένων πανεπιστημιακών, άλλοι προβάλλονται από ερευνητικά κέντρα, άλλοι από διάφορες χώρες μέλη, άλλοι δείκτες προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι οι δείκτες που αναλύονται, η φιλοδοξία τους, αν εφαρμόζεται σε μία ή την άλλη η πολλές χώρες. Βάσει δεδομένων που χρησιμοποιείται υπάρχει συγκεκριμένο κεφάλαιο για το ποιες βάσεις δεδομένων υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη διαμόρφωση των δικτών και τι βελτιώσεις απαιτούνται για να είναι πιο και αυτοί οι δείκτες. Έχουμε μία μεμονωμένη ανάλυση του κάθε δείκτη που υπάρχει στην μελέτη και έχουμε και κάποια συμπεράσματα γενικά. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα. Έχουμε γενικώ αξιόλογους δείκτες που όμως δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικοί. Χρειάζεται λοιπόν ε, περισσότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη συνένεση για τη διαμόρφωση των δικτών, ώστε οι δείκτες αυτοί να χρησιμοποιηθούν ε, κατά την αξιολόγηση ενός ευαίσθητου πολιτικά θέματος, όπως είναι η ποιότητα της εργασίας. Τώρα, κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Ένα από τα προβλήματα των σχολείων είναι ότι στο ίδιο σακί μπερδεύονται μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα εργασίας και απασχόλησης, αλλά και μεταβλητές που σχετίζονται με την ποσότητα, δηλαδή αν ε, δημιουργείται περισσότερη ή λιγότερη απασχόληση. Επίσης υπάρχουν μεταβλητέ που αφορούν την ευημερία του εργαζόμενου ή την ποιότητα μια οικονομία, αλλά δεν συνδέονται άμεσα με την ποιότητα τη απασχόληση. Για παράδειγμα, η παραγωγικότητα, τα συνολικά επίπεδα παιδεία Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά τα γενικά επίπεδα παιδείας, εκπαίδευσης και έχουν θετικό αντίκτυπο στη γενική οικονομία και στην ευημερία, αλλά δεν σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα εργασίας. Θα πρέπει να μετρήσουμε μόνο την ποιότητα εργασίας και εκεί θα δούμε αν χρησιμοποιείται περισσότερη, λιγότερη παιδεία, ε, ειδική, γενική κτλ. Τώρα για την για την ένταση εργασίας. Εκεί λείπουν πολλοί δείκτες. Κάποια στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Μελέτη για την Ποιότητα Εργασίας του Ιδρύματος του Δουβλίνου. Από εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική μεταβλητή της ποιότητας εργασίας που δεν υπάρχει σε άλλους δείκτες. Τις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε, αντί να έχουμε έναν συνολικό δείκτη, ένα σύνολο δικτών. Κάτι τέτοιο δεν μας επιλύει όλα τα προβλήματα. Γιατί στη τελική ανάλυση, όταν έχουμε ένα κατάλογο 15 δικτών, δίνουμε εμείς ως αναγνώστες, ως αναλυτές, δίνουμε περισσότερη σημασία στον έναν ή τον άλλον δίκτυα από τον κατάλογο των 15. Και ουσιαστικά κάνουμε μια ιεράρχηση των δικτών για να βαφθεί το θέμα της στάθμισης και της συνάθρησης, το καλύτερο είναι να έχουμε έναν συνολικό δίκτυ που θα μπορούσε να αναλυθεί, να διαχωριστεί στα επιμέρους του στοιχεία και ο καθένας να διαλέγει το πεδίο σύνθεσης που θέλει. Όταν υπάρχουν τέτοια συνολικά συστήματα, η διακριτική στάθμιση δεν δικαιολογείται. Σε μερικές περιπτώσεις ενσωματώνουμε κάποιους δείκτες ικανοποίησης με την εργασία. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι και πολύ συνεπές, γιατί η ικανοποίηση με την εργασία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Αν εμείς αν μετρήσουμε τα χαρακτηριστικά της εργασίας με άλλους δείκτες, δεν έχει νόημα επιπλέον να βάλουμε και την ικανοποίηση που κανονικά θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο το τμήμα των δικτών είναι ε, δείκτες ε, συνολική αθρηστική, που είναι πολύ πιο εύκολο. Έχουν περισσότερα αθρηστικά στατιστικά στοιχεία από ό,τι μεμονωμένα, αλλά αυτό δεν μας ε, επιτρέπει να καταλάβουμε αν υπάρχει ένα άθροισμα θετικών στοιχείων ή αρνητικών στις ελάχιστες θέσεις εργασίας ή αν ή αν υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των εργασιών που έχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Εδώ μας ενδιαφέρουν περισσότερο ατομικές πληροφορίες και όχι οι Από τις ατομικές πληροφορίες μπορούμε να κάνουμε και μία ανάλυση τη της ποιότητας θέσεων εργασίας, ανάλογα με το φύλλο, με την ε, εθνικότητα και ούτω καθεξής. Παρά τις διαφορές αυτές, όταν αναλύουμε τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από τους διάφορους δείκτες που δημιουργούνται με βάση διαφορετικές προοπτικές υπάρχει μια συνέπεια των αποτελεσμάτων και η κατανομή των χωρών είναι σχετικά λογική, συνεπής. Οπότε με διαφορετικούς τρόπους καταμετρούμε κάτι που ενοιολογικά θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ποιότητα εργασίας που υπάρχει και αντανακλάται με τον, με, τον ένα ή τον άλλο τρόπο στους δείκτες. Οι συντάκτες της μελέτης είναι πεπισμένη ότι έχει νόημα να αφιερώσουμε ενέργεια και χρόνο για να φτιάξουμε ένα δίκτυο ποιότητα εργασία για να καταμετρήσουμε και την καλή συμπεριφορά τη αγορά εργασία που δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, ακόμη και σε περίοδο κρίση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο αριθμό εργαζομένων που έχουν δουλειά, και είναι σημαντικό να ξέρουμε αν αυτή η δουλειά είναι θετική για να αξιολογήσουμε τα κοινωνικά συστήματα και τις πολιτικές απασχόλησης και να δούμε τι είδους απασχόληση είναι αυτή, πώς μεταβάλλεται, τι πολιτικές απασχόλησης ε, υιοθετούνται και πώς επηρεάζουν τον αριθμό των θέσεων εργασία και την ποιότητά τους. Έχουμε και τις τεχνολογικές αλλαγές, έχουμε και την παγκοσμιοποίηση. Εμείς πιστεύουμε ότι οι φυστάμενοι δείκτες δεν ε, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος της περιπλοκότητας και του πολυδιάστατου χαρακτήρα του φαινομένου. Αλλά πιστεύω ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί τέτοιο δείκτης ποιότητας. Μπορώ να κάνω ένα παραλληλισμό με τον τιμάριθμο ή με το δείκτη του ΑΕΠ. Έχουμε τώρα το Labor Force Survey, έχουμε την απογραφή για το εργατικό δυναμικό, έχουμε κάποια στοιχεία και όλοι τα δέχονται. Η δημιουργία των στοιχείων θέσεων απασχόλησης προϋποθέτει μια συμφωνία για το τι εστί εργαζόμενος και τι εστί εργασία. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία για το πώς θα καταμετρήσουμε τις τιμές, να, συμφωνήσουμε για το πώς θα καταμετρήσουμε το ΕΠ. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μιας χρονοβόρας διαδικασίας συζήτησης και συμβιβασμού που κατέληξαν στους δείκτες που έχουμε για το τιμάριθμο, για το ΕΠ και που μπορεί να τροποποιούνται ανεπαίσθητα, αλλά δεν αμφισβητούνται. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα συμβεί και με τον ε, δίκτυ ε, ποιότητας απασχόλησης. Τα προβλήματα που έχουμε με το δίκτυο αυτό είναι παρόντα και σε άλλους δείκτες. Και μερικές φορές έχουμε μια πολιτική ότι όλα χρησιμεύουν και λαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία υπόψη. Αυτό ισχύει όμως και για άλλου δείκτες, όχι μόνο για την ποιότητα εργασία, αλλά και για διάφορε πτυχές της καθημερινότητας. Αυτά και με στη διάθεσή σας για τις απορίες. Ευχαριστώ. Ε, ήταν πολύ χρήσιμα αυτά. Αλλά προτού ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα να πω το εξής ε, θα ήθελα να έχει γίνει περισσότερη εργασία διότι ε, του θέματος γιατί άπαξ έχουμε όλους αυτούς τους δείκτες τι θα γίνει θα μπορέσουν να ενταχθούν στην νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουν να περιληφθούν στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη όταν δηλαδή έχουμε αυτούς τους δείκτες πολλές φορές δεν τους χρησιμοποιούμε δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή καν τις στατιστικές τις οποίες συλλέγουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε πώς σκοπεύετε να τις χρησιμοποιήσετε. Το άλλο θέμα το οποίο αναφέρατε είναι... Ε, ε, δεν, δεν το σχολιάστε όμως τόσο πολύ είναι ε, πώς ε, θα καθορίσουμε την ποιότητα ζωής στο επίπεδο του στρες ε, το οποίο ε, ενδιαφέρει και τους εργαζόμενους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα να υπάρχει ένα σχετικός δείκτης όπως και σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία για το μέλλον, αν είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε ή με άλλους τομείς όπου θεωρείται ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση ή θα πρέπει με τις βέλτιστες πρακτικές να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους. Θα ακούσω όμως δύο ακόμη σχόλια, την Ελίζα Μπεθμωρό και άλλον έναν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή άκουσα την παρέμβαση του συντάκτη της έκθεσης και την δικιά σας, διότι συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία είπατε. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε μία τέτοια εργασία για την εργασία και τους δείκτες θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η χρησιμότητά τους και ε, πώς χρησιμοποιούνται διότι η ποιότητα και η χρήση τους εξαρτάται από την επιστημονική κατάρτιση των ε, δικτών αυτών. Θα πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε για να λάβουμε ε, πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει λοιπόν η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται να βασίζεται σε επιστημονικούς πυλώνες και η δυσκολία στο θέμα αυτό είναι ότι οι δείκτες αυτοί συγχέουν στοιχεία και υποκειμενικά και αντικειμενικά. Άρα θα έπρεπε πρώτον να ξεκαθαριστεί το τοπίο μεταξύ του υποκειμενικού και του αντικειμενικού στοιχείου χωρίς να λέω ότι δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη το υποκειμενικό στοιχείο γιατί αυτή είναι η ε, ανθρώπινη κατανόηση και αντίληψη της εργασίας. Για να μπορέσουμε όμως να τα αντιμετωπίσουμε σωστά θα πρέπει να υπάρχει μια λογική προσέγγιση μεταξύ των δύο πτυχών ιδίως διότι η αντίληψη όπως είπατε στοιχείων τα οποία φαινομενικά είναι αντικειμενικά γίνονται αντιληπτά διαφορετικά και σκέφτομαι την ευελιξία την οποία πολλοί ε, εργαζόμενοι ε, περιμένουν μάλιστα ίσως περισσότερο οι γυναίκες από ότι οι άντρες ε, σε ορισμένες εργασίες, σε ορισμένες ομάδες υπάρχει ε, μία προσμονή μία τακτικής οργάνωσης εργασίας ενώ άλλοι εργαζόμενοι ζητούν διαφορετικά θέματα. Εμείς λοιπόν ε, για να έχουμε μία χρήση πολιτική και αντικειμενική ε, των στοιχείων πρέπει να έχουμε διευκρινίσει και εμβαθύνει τα στοιχεία. Πρέπει να εμβαθύνουμε την επιστημονική μέθοδο κατά τρόπον ώστε να έχουμε μία μέθοδο στην οποία να μπορούμε να βασιστούμε. Και το δεύτερο θέμα στο οποίο ήθελα να παρέμβω ήταν ότι θα χρειαστεί να υπολογίσουμε επακριβώς τις ε, επιπτώσεις της τεχνολογίας της πληροφόρησης στην ποιότητα εργασίας. Αλλάζει κάτι ε, στον τρόπο με τον οποίο η αντιλαμβάνονται τα θέματα τους. Υπάρχει μία ε, αλλαγή για τους ε, ε, για τους εργοδότες και αυτό είναι μεν ενδιαφέρον αλλά χρειάζεται επιστημονική μεθοδολογία για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα σαφή σημεία στην στρατηγική της Λισαβόνας περιμένουμε μία ανάταση και μία καλύτερη ποιότητα εργασίας για να οδηγηθούμε όμως προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε καθηγητά Ραφαέλ Μουνιός Δεμπουστίγιο. Είχα την ε, ευκαιρία να διαβάσω και μία από τις μελέτες σας, αλλά με τη ζωντανή παρουσίαση κερδίζετε ακόμη περισσότερο και ελπίζω να μην είναι η τελευταία φορά που σας βλέπουμε, γιατί βρισκόμαστε στην αρχή μίας ε, μακράς πορείας. Λέτε στο τέλος της μελέτης σας ότι θα πρέπει να υπάρχει μία διπλή προσέγγιση μια προσέγγιση επιστημονικής συνένεσης και ταυτόχρονα μιας, ε, μια πολιτικοκοινωνική προσέγγιση για την διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος. Από ακαδημαϊκή και επιστημονική άποψη υπάρχει αυτή η σύγκληση μεταξύ των ερευνητών, μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων. Γιατί θα ήταν χρήσιμο για μας τους πολιτικούς να γίνει μια προεργασία σε ένα τόσο δύσκολο έδαφος, ε, γεμάτο ερωτηματικά και τόσο πολύ σύνθετο και πολύ διάστατο. Και πριν λάβουμε την πολιτική απόφαση είναι χρήσιμο να έχουμε εμπεριστατωμένη και έγκυρη ενημέρωση για τις διάφορες πτυχές αυτού του πολυδιάστατου ζητήματος. Όπως είπε και η Ελίζαμπεθ, αυτή τη στιγμή ζητούμε το δεύτερο τμήμα της διαδικασίας της Λισαβόνας να δώσει έμφαση στα θέματα ποιότητας. Χθες είχαμε συνεδρίασή μας στον Επίτροπο Αλμούνια και εκεί βλέπω ότι μόνο μια ποσοτική αξιολόγηση της ε, εργασίας δημιουργεί κακής ποιότητας, ε, κακής παραγωγικότητας ε, θέσεις εργασίας και πολύ ευάλωτες και δεν ε, δίνει αρκετά εφόδια στον κόσμο να αντέξει την πρώτη καταιγίδα. Όπως ε, συνέβη στην Ισπανία που χάθηκαν ε, πολύ γρήγορα θέσεις απασχόλησης που χρειάστηκε 10 χρόνια για να δημιουργηθούν. Σας ερωτώ λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε, ποια είναι η δική σας γνώμη και πώς θα μπορούσαμε και εμείς να συμβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πλαισιώσουμε αυτήν την κοινωνιολογική έρευνα. Γιατί αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερευνητική κατεύθυνση και εκεί θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πόρους στα ερευνητικά κέντρα, στα κέντρα μελετών και στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για να προχωρήσουν και να βαθύνουν αυτό το είδος τη μελέτη. Έχω και μια άλλη ακαδημαϊκή ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι συμμετέχουμε στο παγκόσμιο όραμα της αξιοπρεπούς εργασίας υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και έχουμε και κάποιες ε, παγκόσμιες αλλαγές. Μήπως πιστεύετε θα πρέπει να τροποποιήσουμε τους δείκτες ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Μήπως θα πρέπει να θετήσουμε μια ευρωπαϊκή ερμηνεία για τους δείκτες αυτούς. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, μήπως είναι αντιφατικό. Είναι σκόπιμο να έχω μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για το πώς αντιμετωπίζουμε την ποιότητα εργασίας ε, στην ε, Ευρώπη σε σχέση με τις προδιαγραφές ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εργασία. Σας ευχαριστώ. Πριν ε, ε, συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, να δώσω το λόγο στον ομιλητή να απαντήσει. Αν συγγνώμη, να ακούσουμε μια ερώτηση ακόμα από την κυρία Στρέντερ. Η ερώτησή μου είναι η εξής, στην ίδια κατεύθυνση όπως και ο συνάδελφος Σέρκας, ο οποίος είπε ότι ε, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι ε, πώς διεξάγονται οι ε, διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας της μελέτης σας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, ποια από τα κριτήρια και τα μέτρα εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας ε, στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής απασχόλησης και τι ε, μέτρα έχετε λάβει ε, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, μία σύσταση η οποία είναι χαμηλότερο επίπεδο. Δεν βλέπω να υπάρχει μια τέτοια ταξινόμηση και ε, αν προχωρήσουμε όπως ε, εσείς ε, προτείνετε θα χρειαστεί μια ευρωπαϊκή νομοθετική εργασία δηλαδή θα πρέπει τα πρότυπα να αναμορφωθούν βάσει της ανάλυσής σας και θα σας παρακαλούσα να διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Εάν θέλετε να απαντήσετε σε αυτά τα τέσσερα ερωτήματα και μετά θα υπάρξουν άλλα τέσσερα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και μάλιστα ορισμένα από τα θέματα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα οπότε θα προσπαθήσω να τα απαντήσω συνολικά. Ε, καταρχήν, γιατί να καταρτήσουμε έναν δείκτη ε, ποιότητος ε, της απασχόλησης σαν κοινωνιολόγος για μένα αυτό είναι σαφές αλλά για την ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να τεθεί το θέμα αυτό και επανέρχομαι εις ε, τους όρους οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν δηλαδή ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί δεν υπάρχει και πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει ε, και από μία αρχή της στρατηγικής της Λισαβόνας ε, το 2005 σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θέμα αυτό δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή χρειάζεται καλύτερη και περισσότερη απασχόληση αλλά μπορούμε να μετρήσουμε το ποιοτικό, όχι όμως το το ποσοτικό όχι όμως το ποιοτικό και αναρωτιόμαστε στην Ισπανία αν οι θέσεις εργασίες που δημιουργούνται είναι καλής ποιότητας και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μπορώ έμεσα να απαντήσω βασιζόμενος ή στην παραγωγικότητα και στο είδος του συμβολέου. Αλλά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο δίκτυο ενώ μπορώ ποσοτικά να σας πω ακριβώς πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν χωρίς να μπορώ να σας πω αν οι θέσεις αυτές είναι ποιοτικέ και αν ε, ε, έχουμε ε, απασχολήσεις χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν λοιπόν τα, τα ακραία αλλά εγώ δεν έχω δείκτες για να μετρήσω το κέντρο. Υπάρχει μία μία συνενετική βάση ε, η οποία βασίζεται ε, σε, ε, σε κοινωνική προσέγγιση και όχι επιστημονική και θα μπορούσα να ελέγξω τις θέσεις οι οποίες δημιουργήσαν στην Ισπανία μετά την ύφεση. Επίσης να δούμε πώς επηρεάζει η κρίση την ποιότητα της απασχόλησης σε ό,τι αφορά το στρες. Η κρίση επιτείνει το άγχος των ε, εργαζομένων. Δεν έχουμε τέτοιους δείκτες για να μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση. Και αν θεωρούμε ότι η ποιότητα της εργασίας είναι μια μεταβλητή, ένα στοιχείο που χρήζει της προσοχής μας, αξίζει της ε, προσοχής μας και της ανησυχίας μας. Αν μας ανησυχεί λοιπόν, να μας προβληματίζει αυτό το θέμα της ποιότητας της απασχόλησης, για να μην είναι πια μόνο ένα θέμα προγραμματικών δηλώσεων. Χρειαζόμαστε, αν όντως μας προβληματίζει αυτό το θέμα, ένα δείκτη για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτή την ποιότητα εργασίας. Ένας τέτοιος δείκτης θα μας χρησίμευε να δούμε αν υπάρχει συνδυασμός θετικών και αρνητικών στοιχείων σε μια δεδομένη εργασία αν υπάρχει αντιστάθμιση. Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε σήμερα. Η κυρία Πρόεδρο μίλησε για το άγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το θέμα του στρε, του άγχου. Και το, θέμα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο δίκτυο. Και μπορούμε να έχουμε και παραδείγματα για αυτό το ανοιχτό μοντέλο δικτών. Γιατί εκεί υπάρχουν κάποιοι δείκτες με συγκεκριμένα παραδείγματα για το άγχος όπως μας δείχνει η μελέτη για την ποιότητα εργασία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο. Αλλά εκτό από το άγχο, έχουμε και άλλα αρνητικά στοιχεία. Μήπω όμω υπάρχουν αντισταθμίσει με θετικά στοιχεία, ώστε σε τελική ανάλυση το έργο του Ευρωβουλευτή να μην είναι, κακή, να μην είναι κακής ποιότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια συνολική άποψη και να μην ε, επικεντρωθούμε σε ένα και μόνο σημείο. Τώρα, από τη στιγμή που θα κατασκευάσουμε, που θα φτιάξουμε αυτό το δίκτυο, τι πολιτικό αντίκτυπο θα έχει. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ να μπω στη δική σας θέση, εκτός και αν εκλεγώ ευρωβουλευτή την επόμενη φορά και τότε θα προτείνω εγώ ή θα συμμετέχω στη λήψη μιας απόφασης. Εγώ πάντως πιστεύω ότι χωρίς σωστή ενημέρωση δεν μπορεί κανείς να λάβει εμπεριστατωμένα μια απόφαση. Και η απόφαση είναι αν θα γίνει παρέμβαση ή όχι και σε τι τομέα, στο τομέα της, του συντονισμού, στο τομέα των βέλτιστων πρακτικών, σε τομέα υποδείξεων, συστάσεων, σε νομοθετικό επίπεδο, ρυθμιστικό και κανονιστικό. Για να λάβει κανείς μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να έχει συλλέξει αρκετά στοιχεία, να έχει αρκετή γνώση της πραγματικότητας, ε, ώστε να μπορέσει να λάβει μια εμπεριστατωμένη γνώμη και απόφαση. Και στην τελευταία ερώτηση, για το κατά πόσο θα πρέπει να καταλήξουμε σε ελάχιστους κανόνες, ποιος είμαι εγώ για να πω κάτι τέτοιο. αυτή θα μπορούσε να είναι η προσωπική μου γνώμη, αλλά εδώ αυτή η γνώμη ως προσωπική γνώμη δεν αξίζει τίποτα. Είναι η γνώμη ενός απλού Ευρωπαίου πολίτη. Ως επιστήμονας πάντως, κοινωνικών επιστημών, για να πούμε αν χρειαζόμαστε ελάχιστους κανόνες θα πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε την ποικιλομορφία της ποιότητας εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν αυτή η ποικιλομορφία μας σκανδαλίζει ως Ευρωβουλευτές, τότε ίσως χρειαστεί να λάβουμε μία απόφαση μετά από συζήτηση για το κατά πόσο χρειάζονται ελάχιστοι κανόνες. Πάντως, από ό,τι φαίνεται από άλλους τομείς σε κοινωνικά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ τη παρέμβαση και τη επιβολή ελάχιστων κανόνων. Και δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο στην απασχόληση, ενώ δεν έχει γίνει σε άλλου τομεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαξιώνεται ο δείκτη τη ποιότητα. Γιατί οποιαδήποτε γνώση μα είναι χρήσιμη. Και αν τώρα κάναμε μια ψηφοφορία ρωτώντας ποιοι πιστεύουν ότι στην Ευρώπη η απασχόληση επιδεινώθηκε με την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών ή με την κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών τα τελευταία 20 χρόνια. Ποιοι πιστεύουν ότι επιδεινώθηκε η απασχόληση και ποιοι θεωρούν ότι βελτιώθηκε. Δεν μπορώ να γνωρίζω το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία. Αλλά και η ομοφωνία να υπάρχει, αυτή στηρίζεται σε πεπιθήσεις. Εγώ σας λέω ότι ασχολούμαι με το θέμα αυτό 10 ώρες τη μέρα. Αλλά όταν κληθώ να απαντήσω, περισσότερο θα εμπιστευτώ το ένστικτό μου, γιατί πραγματικά αδιάσυστα στοιχεία δεν υπάρχουν. Δεν είναι σαφές αν βελτιώθηκε ή όχι η εργασία, αν επιδεινώθηκε. Σε ορισμένες χώρες φαίνεται επιδεινώθηκε, σε άλλες χώρες βελτιώθηκε, σε άλλες χώρες υπάρχουν ασύμετρες βελτιώσεις, σε ορισμένες υπάρχει πόλωση. Γι' αυτό και όσο περισσότερο επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία, τόσο πιο βαθιά φτάνουμε στο, στο φαινόμενο αυτό. Τώρα για το κατά πόσο υπάρχει συνένεση στη βιβλιογραφία. Η κοινωνιολογία έχει μεγαλύτερη εμβάθυνση στο θέμα αυτό από το Μάρξ και από όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την κοινωνιολογία της εργασίας. Τώρα, η οικονομία θεώρησε ότι υπήρξαν αντισταθμίσεις και μπορεί κάποιες κακές προϋποθέσεις, συνθήκες εργασίας με καλύτερο μισθό υπάρχει αντιστάθμιση. Αλλά αυτό συμβαίνει σε μια ιδεατή αγορά. Αλλά η αγορά εργασία δεν είναι ιδανική, οπότε η θεωρία της αντιστάθμισης του Άνταμ Σμιθ, που πρωτοϋποβλήθηκε πριν από 200 χρόνια, δεν εφαρμόζεται πάντα τουλάχιστον. Εκεί όμως που σημειώνεται πρόοδος και φαίνεται στο δεύτερο ή τρίτο κεφάλαιο της μελέτης, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν είναι πανεπιστημιακή μελέτη, είναι αν εξιολογείται πολυδιάστατος χαρακτήρας της ποιότητας εργασίας και η σημασία των τομέων που έλυθησαν υπόψη. Στην γραφική παράσταση που σας έδειξα, βλέπω, είδαμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία σύνεσης. Παρακολουθώντας και την βιβλιογραφία για την κοινωνιολογία. Ο καθηγητή Φράνσις Γκριν και άλλοι που μίλησαν για το θέμα αυτό λένε πάνω κάτω αυτό που λέμε και εμεί στη μελέτη. Υπάρχει μια συνένεση ω προ την πρόπτικη. Υπάρχει αρκετή συνένεση λοιπόν για να εμβαθύνουμε τις εργασίες για την κατασκευή ενός δίκτυ. Τώρα αν θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε με, τη, με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, εγώ πιστεύω ότι ναι, θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες γιατί η πολιτική και το πρόγραμμα της αξιοπρεπούς εργασίας του Decent Work ε, πιστεύω θα πρέπει να το συμμεριστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί και ένας ειδικός δείκτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μια καλή ή μια κακή εργασία δεν είναι άσχετη με το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας. Και ένας από τους λόγους που σας επισήμανα στη μελέτη και το παρέλειψα στην παρουσίαση είναι ανάλογα με την ε, εξέλιξη, την ανάπτυξη μιας χώρας ε, γινόμαστε και πιο απαιτητικοί για, ως προς την απασχόληση και αυξάνεται και η ελαστικότητα. Σε μια κοινωνία που, σαν τη δική μας που μεταβάλλεται, το θέμα της ισορροπίας των φύλων είναι πολύ σημαντικό. Πριν από 30-40 ε, χρόνια στην ε, Ισπανία δεν ήταν σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί οι γυναίκες δεν δούλευαν πριν από 30-40 χρόνια. Τώρα όμως που οι γυναίκες έχουν ενταχθεί στο χώρο εργασίας, στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να λυθεί και αυτό το στοιχείο υπόψη στις μελέτες. Κάτι που ισχύει για μας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι ακόμη για τη Μαυριτανία, για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο Είναι κάπως διαφορετικό από το πρόγραμμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ή του ΟΗΕ, της ΠΝΙΤ, για το δίκτυ ανάπτυξης του ανθρώπου, αλλά για, την, για τη φτώχεια, για το δίκτυ της φτώχειας, έχουμε ένα δίκτυ για το ποσοστό φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και άλλο δίκτυ για το ποσοστό φτώχειας στις ανεπτυγμένες χώρες. Τώρα το να αισθενιστούμε το πρόγραμμα Decent Work και αυτό κάπως προβληματικό είναι γιατί δεν υπάρχει ένας και, μόνος, ένας και μόνο δείκτης. Υπάρχει μια έννοια που μπορεί να αντανακλαστεί σε 4-5 διαφορετικούς δείκτες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός δίκτυ. Ίσως θα έπρεπε να είναι πιο φιδωλός, να έχει λιγότερες μεταβλητές, γιατί οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες ε, έχουν και λιγότερο ανεπτυγμένα στατιστικά συστήματα. Οπότε αν θέλουμε ένα ε, εφικτό και εφαρμόσιμο δίκτυ θα πρέπει να είναι λιγότερο φιλόδοξος. Πάντως εμείς έχουμε καλές στατιστικές και μπορούμε να τις προχωρήσουμε. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ε, αξίζει τον κόπο να αφιερωθούν πόροι και ενέργεια για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δίκτυ ποιότητας. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και βασικό στοιχείο της στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα. Η διαμόρφωση ενό δίκτυ, αν θέλουμε να ληφθεί υπόψη σοβαρά το θέμα της ποιότητας της εργασία. Και αυτό είναι ένα βήμα που θα πρέπει να γίνει εδώ και όχι σε ένα ερευνητικό κέντρο, αλλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Yes, thank you. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη ώρα, γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση μετά τις 11 ε, και 4. Αλλά έχουμε ακόμη πέντε ομιλητές στον κατάλογο. Να τους ακούσουμε και μετά να ακούσουμε και τις απαντήσεις σας για να ολοκληρώσετε. Η κυρία Πλάμ. Σας ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ραφαριμούνιος και θα ήθελα να προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να μην επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, τα οποία υποστηρίζω απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, εξηγήσεις που μας ε, δώσατε. Νομίζω ότι αυτή, αυτό το νέο σύστημα που προτείνεται, αυτοί οι δείκτες με τους οποίους μετράτε η ποιότητα της εργασίας αποτελούν μία πρόοδο. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της ποσόστοσης των εργασία της εργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις γυναίκες και αυτό αποτελεί σημαντικό στόχο για μας. Και πέρα από τη συμμετοχή των γυναικών στην ε, στο χώρο εργασίας τίθεται και το θέμα της ποιότητας των, της εργασίας των γυναικών και θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι υπάρχει ακόμα διαφορά μισθού ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Με τους δείκτες αυτούς που συντάσσεται για την ε, ποιότητα της εργασίας και στις πολιτικές που καταρτίζουμε προκειμένου να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα των μισθών και να υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην ε, αγορά εργασίας. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι σχετίζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ραστή. Ράπτη. Oh, sorry. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Καθηγητά, ευχαριστώ για τις ε, πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε μέσα από τη μελέτη σας και θέλω να ρωτήσω πάρα πολύ σύντομα τρία πράγματα. Ε, μάλλον δύο. Το ένα είναι η αναφορά που κάνατε στην αξιοπρεπή εργασία. Decent work είναι ένας όρος που ιδιαίτερα σε χώρες που υπολείπονται σε νομικό πλαίσιο, σε νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τα ζητήματα απασχόλησης και εργασίας, ε, το decent work είναι μια πολύ ευρία έννοια. Ε, θα ήθελα, εάν μπορείτε, να μας πείτε α, κάποιο κάποιους πιο συγκεκριμένους παράγοντες και στοιχεία που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την αξιοπρεπή, τον όρο αξιοπρεπή εργασία. Και το δεύτερο και τρίτο μαζί είναι το εξής. Ε, βλέποντας εδώ τη μελέτη σας, ε, πηγαίνω σε δύο α, χάρτες. Ε, ο ένας είναι στη σελίδα 35 και αφορά, είναι Index of ε, Job Satisfaction και ο άλλος είναι στη σελίδα 41, αφορά το percentage of people who would enjoy having a pet job even if they did not need the money. Βλέπω, μάλλον δεν βλέπω σε αυτά τα δύο ιστογράμματα να υπάρχουν δύο χώρες του Νότου, η Ιταλία και η Ελλάδα. Ε, συμπτωματικά δεν είναι δύο από τις πέντε χώρες που, για τις οποίες χτες ο κύριος Αλμούνια ανέφερε ότι βρίσκονται στο κόκκινο στα ζητήματα απασχόλησης και σχέσεις με τα δημοσιοοικονομικά. Ρωτώ λοιπόν, το γεγονός ότι δύο αυτές χώρες λείπουν από το είναι απλά γιατί δεν υπήρξαν στοιχεία ή για κάποιους άλλους λόγους. Ε, κλείνω και σας ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες. Thank you. Uh, σας ευχαριστώ. Κυρία σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το κατά πόσο υπάρχει ε, ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την ε, εργασία. Φυσικά είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες. Στις ε, σκανδιναβικές ε, χώρες και αντίδρα στη Φιλανδία εξετάζουμε αυτό το παράγοντα επί σειρά ετών και προσέξαμε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά συνδικάτα και παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων ε, στην ε, εργασία, πολλοί αντικειμενικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι θετικοί λοιπόν, αποδεικνύεται ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να ακολουθήσει κανείς ε, μία σταδιοδρομία Συνήθως η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 58-59 έτη. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η αιτία αυτής της ε, πρόορης συνταξιοδότησης. Υπάρχει κάποια κόπωση, υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, υπάρχει ε, παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Κατά ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η εργασία των προϊσταμένων μπορεί να εξελιχθεί. Μπορούν να υπάρξουν διαφορετικοί δείκτες για να καταμετρηθεί αυτή η διάσταση και γενικά ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν οι θέσεις εργασίας. Άτομα τα οποία μένουν στην ίδια θέση για δεκαετίες είναι σπάνια. Οι πιο πολλοί έχουν πλέον επισφαλείς θέσεις εργασίας και αυτή η γενική τάση αλλαγής πώς επηρεάζει το πόσο ικανοποιημένος είναι ο κόσμος από τη δουλειά του. Και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες προσέχουμε ότι πολλοί εμπειρογνώμονες δεν μπορούν να διαχωρίσουν πλέον τον χρόνο εργασίας από τον ελεύθερο χρόνο τους. Γιατί συχνά εργάζονται και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους χρειάζεται κανείς για παράδειγμα να είναι συνδεδεμένος με το ίντερνετ, να κοιτάει τα email του ακόμα και όταν είναι ε, στον ελεύθερο χρόνο του. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Διακνέρη, ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Κύριε Δημοστήγιο, Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, για την Επιτροπή μας, γιατί είναι και αν θέλετε η άλλη πλευρά του νομίσματος της χρηματοοικονομικής κρίσης. Ε, ξέρω πώς είναι η εργασιακή κατάσταση στην Αυστρία και το σχετικό σου δείκτης εργασιακής ατμόσφαιρας που προσπαθούμε να, να αναπτύξουμε σε εθνικό επίπεδο. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, πολύ καλές ε, εθνικοί όροι εργασίας. και θα έπρεπε να τεθεί, αν θέλετε, το θέμα των, ευρω... δικτών ε, εργασίας σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή στο ΙΜΠΕΡ για την καλύτερη νομοθεσία. Ξέρω ότι το θέμα αυτό της αξιολόγησης της θέσης εργασίας ε, είναι, αν θέλετε, άλλη μια διάσταση και θα ήθελα να διευκρινίσω και την ερώτηση της κυρίας Σρόιντερ. Θεωρείτε ότι σε κάποια ορισμένη χρονική στιγμή θα πρέπει να είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ε, κατάλληλα μέτρα, μια κοινή ομάδα δικτών όπου θα συμπεριληφθούν πολλοί, πολλές διαστάσεις γιατί νομίζω ότι ο χρονικός παράγοντας είναι και αυτός μια διάσταση την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση να απευθύνω στον καθηγητή για τους δείκτες. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνος δείκτης. Μία δυνατότητα θα ήταν να πούμε ότι η ομοφωνία αυτή ε, προέρχεται από τις ρυθμίσεις των κοινωνικών ε, εταίρων. Αυτό είναι το ένα κριτήριο. Επίσης, στις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει αυτή η άμεση σχέση μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό το ξέρουμε και κάποιοι λένε ότι ο παράγοντας ε, σταθεροποίησης είναι ένα ελάχιστο εισόδημα, δηλαδή ε, μια οικονομική δικλίδα. Να κοιτάξουμε για παράδειγμα το παράδειγμα της Opel, γιατί με απασχολεί το θέμα αυτό, είναι στην εκλογική μου επιφέρεια. Το τελευταίο χρόνο μάθαμε πάρα πολλά για την ικανοποίηση από την ε, εργασία για υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους. Μιλάμε για ένα προϊόν ή περισσότερα προϊόντα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν στην αγορά. Πριν από κάποια χρόνια θα έλεγα ότι πολύ ωραία είναι πάρα πολύ περήφανοι όσοι εργάζονται στην εταιρεία αυτή. Αυτό είναι το τμήμα της ικανοποίησης ε, από την εργασία τον οποίο χρειάζομαι. Ναι, μεν υπάρχει το στρες, αλλά το αποδεχόμαστε γιατί υπάρχει μελλοντική διάσταση. Τα ίδια άτομα όμως σε μια κατάσταση όπως η σημερινή, όπου διαπιστώνει η General Motors ότι α, θα κρατήσουμε την όπολη και δεν πρόκειται να την πουλήσουμε και έχουμε ένα χρόνο ε, τρομακτικών αναταραχών ε, στοιχήσαμε πάρα πολλά χρήματα φορολογουμένων, αλλά σήμερα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτω ικανοποίηση από την εργασία, γιατί υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει μελλοντική διάσταση πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να διατυπωθεί ένας άλλος δείκτη, προκειμένου να υπάρχει μια σταθεροποίηση της ε, κοινωνία μα να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια κουλτούρα των επιχειρήσεων, χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα διατυπώσουν μια αρχή και την οποία θα διατηρήσουν στη συνέχεια. Χρειαζόμαστε κάτι με το οποίο θα, στο οποίο θα συμμετάσχουμε, να υπάρχει μια μελλοντική διάσταση. Γιατί, αν θέλετε, και οι διευθυντέ μπορούν να φύγουν και θα του απασχολεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτοί που εργάζονται στην επιχείρηση δεν πρέπει κάτι να του δώσουμε ω ε, δικλίδα. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την επιχείρηση να δώσει κάτι, αλλά ίσω θα μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα για να βετεποθεί και να καθιερωθεί μια επιχειρησιακή κουλτούρα και ε, ένα κλίμα υπευθυνότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι η πολιτική μας ε, ε, το πολιτικό μας καθήκον και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον δίκτυο τον, που, το συνετικό τον οποίο αναφέρατε. Um, πέντε λεπτά για να απαντήσετε αν θέλετε. Ξέρω ότι θα δυσκολευτείτε πολύ να απαντήσετε σε πέντε λεπτά, αλλά αν μπορείτε. Ε, Ευτυχώς πολλές από τις ερωτήσεις έχουν ένα κοινό στοιχείο και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε ευθύ εξ αρχής. Ένας δείκτης ποιότητας απασχόλησης δεν είναι δείκτης ικανοποίησης με την εργασία. Τουλάχιστον κατά τη δική μας γνώμη των συντακτών της μελέτης. Αν μπορούσαμε να καταμετρήσουμε την ποιότητα της απασχόλησης με βάση μόνο την ικανοποίηση της εργασίας, ε, θα γινόταν αυτό. Υπάρχουν δείκτες ικανοποίησης με την εργασία και συνολική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σφαιρική, αλλά και ειδική για κάθε χώρα. Κάθε χώρα έχει έρευνες για τις συνθήκες εργασίας και υπάρχουν ερωτήσεις για την ικανοποίηση. Αυτό θα ήταν απλό άμα ταυτιζόταν τα δύο πράγματα. Μετά όμως την ε, μελέτη της συμπεριφοράς των δικτών το επιτελείο μου έφτασε στο συμπέρασμα ότι δεν μας εξυπηρετούν αυτοί οι δείκτες. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένος, πανευτυχής με την εργασία του, παρόλο που αντικειμενικά η δουλειά του είναι αξιολύπητη, είναι κακής ποιότητας. Υπάρχουν μεμονωμένοι οι ατομικοί μηχανισμοί προσαρμογής των προσδοκιών που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το παράδοξο. Κάποιος είναι ικανοποιημένος με μια δουλειά που είναι χάλια. Και Υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν τέτοιες, τέτοιους δείκτες ικανοποίησης και παρόλα αυτά οι προδιαγραφές εργασίες δεν πληρούν καν τα, τους ελάχιστους κανόνες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ας μη συγχαίουμε λοιπόν την ικανοποίηση από τη δουλειά με την ποιότητα της απασχόλησης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί για την ικανοποίηση έχουμε μια υποκειμενική αντίληψη. Κάποιος μπορεί να έχει μια καταπληκτική δουλειά και επειδή δεν προσαρμόζεται στις φιλοδοξίες του, στις προσδοκίες του, να, τη θεω... να μην είναι ικανοποιημένο. Μπορεί να έχει ελαστικό ωράριο, μπορεί να έχει υλικές προϋποθέσεις, καλό μισθό. Αλλά επειδή έχει πρόβλημα στη σχέση του με τον προϊστάμενο, επειδή ε, χρειάζεται να μετακινηθεί πολλή ώρα για να πάει στη δουλειά του, μπορεί να τον δυσαρεστεί η δουλειά του. Αυτό όμως δεν είναι θέμα ποιότητας της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, αλλά διαφοράς μεταξύ των συγκεκριμένων φιλοδοξιών του συγκεκριμένου εργαζόμενου. Η δουλειά είναι καλή, αλλά δεν υπάρχει συντέργεσμα το, τη συγκεκριμένη θέση εργασία με τι ανάγκε του συγκεκριμένου εργαζόμενου. Γι' αυτό λέω ότι δεν ταυτίζονται ικανοποίηση και ποιότητα απασχόληση. Και παραλαμβάνω, υπάρχουν ήδη δείκτε ικανοποίηση από την εργασία. Και αν υπάρχει ένα δείκτη, σίγουρα υπάρχει και ένα οικονο... οικονομολόγο, ένα οικονομέτρη, ένα ε, στατιστικολόγος που εκπονεί όλα αυτά τα στοιχεία, τα συγκεντρώνει και τα αναλύει. Αλλά η ποιότητα της εργασίας είναι μια μεταβλητή που δεν έχει καταμετρηθεί ακόμα, γιατί δεν υπάρχει ειδικό δείκτης. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα περάσουμε από αντικειμενικά χαρακτηριστικά, παρόλο που μερικές φορές καταμετρούνται ε, υποκειμενικά, για το επίπεδο του άγχους πρέπει να το ρωτήσουμε από κάποιον. Αν υπάρχει παρενόχληση, εργασία και αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εργαζόμενο και η αντίληψη του μπορεί να είναι υποκειμενική. Δεν υπάρχει αντικειμενικός δείκτης για την καταμέτρηση της παρενόχλησης, για παράδειγμα, ή του άγχους. Παρόλο που ο δείκτης λοιπόν είναι υποκειμενικός, είναι μεροληπτικός, για να προσεγγίσουμε κάποια στοιχεία και να καταλήξουμε σε αντικειμενικούς δείκτες, λαμβάνουμε υπόψη και κάποιους, ε, κάποιες υποκειμενικές ε, αναλύσεις. Κάποιοι μου είπαν για τη Σουηδία το θέμα της απασχόλησης, εργασίας και της αναψυχής, της ψυχαγωγίας. Και εκεί είναι διαπερατά τα όρια. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε, να βρούμε κάποιους τρόπους να περιλάβουμε και αυτό το θέμα στους δείκτες. Αλλά επανέρχομαι στην ερώτηση του τελευταίου ομιλητή. Ο πατέρας μου που πολύ θα χαιρόταν αν ήξερα ότι τον αναφέρω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έλεγε συνέχεια την ε, Ισπανική παροιμία που λέει ότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Δηλαδή, δεν θα πρέπει από τη στιγμή που δεν έχουμε κανέναν δείκτη να θέλουμε ένα δείκτη που θα τα αναλύει όλα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, θα είναι τέλειος να μην είμαστε του ή όλα ή τίποτα. Από τους δείκτες θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δεν μπορούν να μας καλύψουν όλες τις ανάγκες μας. Όταν έχουμε το δείκτη του ΑΕΠ δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως δείκτη ευημερία. Ο δείκτης του ΑΕΠ μετράει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Δεν μετράει την ευημερία. Αν ζητούμε από ένα δείκτη κάτι για το οποίο δεν είναι προγραμματισμένος, του αναχρηστεύουμε ουσιαστικά. Το θέμα της συμμετοχής σε μια επιχείρηση, του ανήκειν στην επιχείρηση, είναι ζήτημα άλλου δείκτη. Και η συμμετοχή είναι πολύ σημαντική σε μια επιχείρηση. Να έχει ο εργαζόμενος την αίσθηση ότι μετράει στην επιχείρηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι ένα άλλο πεδίο που καλύπτεται στο γενικό μοντέλο. Τώρα, συμμετοχή με ποιο τρόπο, μέσω των συνδικάτων, άμεση συμμετοχή στις μικρές επιχειρήσεις, πώς θα ποσοτικοποιηθεί αυτή η συμμετοχή. Και τη στιγμή που διαμορφώνουμε ένα δίκτυ, υπάρχει, βλέπουμε μια πολύ σημαντική διάσταση για την ποιότητα εργασία, αλλά δεν υπάρχει σαφή μεταβλητή. Ε, σε τέτοια περίπτωση εγκαταλείπουμε αυτή τη μεταβλητή. Καλύτερα να αφήσουμε έξω ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε, να το καταμετρήσουμε σωστά, παρά να το συμπεριλάβουμε και να μολύνει, να παξιώσει τελικά τον ίδιο το δίκτυ. Να δούμε τι μπορούμε να καταμετρήσουμε και τι, μπορούμε, και τι δεν γίνεται να καταμετρηθεί. Επίσης, ε, πόσες μεταβλητές θα συμπεριλάβουμε, πολλές ή λίγες. Δεν είναι το θέμα της ποσότητας των μεταβλητών, νομίζω, το πιο σημαντικό. Και όσο πιο λίγες είναι οι μεταβλητές, τόσο πιο διαφανής είναι ο τρόπος εργασίας. Και η διαφάνεια μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε τι καταμετρούμε, με ποιο τρόπο το μετρούμε και πώς γίνεται η στάθμιση των διαφόρων μεταβλητών. Υπάρχουν μέθοδοι για να περιλάβουμε τομείς όπως ε, αν κανεί εργάζεται με βραχύτατε προθεσμίε και άρα με μεγαλύτερη πίεση ή μπορεί να έχουμε 4-5 μεταβλητέ και με αυτέ τι 4-5 μεταβλητέ να διαμορφώσουμε μια θρηστική μεταβλητή και να περιορίσουμε το πεδίο των μεταβλητών. Τώρα αν θα βάλουμε περισσότερα ή λιγότερα, χάρη στου υπολογιστέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε να προσθέσουμε όσα στοιχεία θέλουμε. Αλλά να προσθέσουμε τι σωστέ μεταβλητέ. Γιατί οι μερικοί δείκτες έχουν 100 και μεταβλητέ και επειδή είναι το ίδιο να έχουμε 50 ή 100, τις προσθέτουμε όλες. Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Τώρα, ο χρόνος. Ο επιστημονικός εντός εισαγωγικών χρόνος μπορεί να είναι σύντομος. Ένας χρόνος, για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει και ο χρόνος της συζήτησης. Και όταν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση, δεν εννοώ ότι θα συμφωνήσουμε όλοι μεταξύ μας. Ε, να είμαστε ενδοτικοί. Θες αυτό το προσθέτουμε, θες εκείνο το προσθέτουμε. Να ειστηρίζεται σε επιστημονική βάση. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει ο, ο δείκτης και θα συζητηθεί, όλοι θα πρέπει να τον υποστηρίξουν για να μην είναι ένας επιπλέον δείκτης χωρίς αξία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των φύλων, ένας δείκτης σαν αυτό που προτείνουμε στη μελέτη δεν μας επιτρέπει επιτρέπει να μάθουμε το χάσμα το μισθολογικό. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Αλλά θα ξέρουμε οι θέσει εργασία των γυναικών τι συνθήκες έχουν ως προς τους μισθούς, την ελαστικότητα, τις δυνατότητες προαγωγής, τις φυσικές συνθήκες κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά εξαιρετική η απάντησή σας. Ακούσαμε με ενδιαφέρουν όσο μας είπατε και αναμένουμε με ανεπομονησία τις υπόλοιπες εργασίες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η βελτίωση της ε, ε, εργασίας και έχουμε την ε, εισηγήτρια. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, Πρέπει να σας πω ότι ελπίζω ότι εφόσον υιοθετήσαμε την έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγγύων λεχονών και γαλακτου και εργαζομένων που θελεάσουν. Ε, θέλω να στηρίξω την πρόταση της ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζει την θέση των εγγύων και λεχώνων αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε με τροπολογίες το κείμενο που έχει καταρτιστεί και επίσης να προσθέσουμε τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει οι κοινωνικοί εταίροι διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν καλύτερα να συμβιβάσουν την εργασία την οικογένεια και να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι χρειαζόμαστε μία πιο ε, σημαντική ε, συμμετοχή των ε, γυναικών στην αγορά εργασίας ε, για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα ανά τον κόσμο. Γι' αυτό και όταν θα συζητήσουμε το θέμα αυτό πρέπει να θεωρήσουμε ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για να υπερβούμε την οικονομική κρίση, να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσουμε ε, τη σχέση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής γονής προωθώντας την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και ένα βασικό θέμα είναι η παράταση της, ε, ε, της αδείας ε, ε, κατόπιν του τοκετού με βελτίωση το, της αποζημιώσεως κατά την περίοδο αυτή. Όσον αφορά την παράταση ε, το, της αδείας τοκετού θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να επιτρέψουμε στις γυναίκες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους αλλά και στην εργασία τους διότι όταν οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν τότε υπάρχει και μεγαλύτερη γονιμότητα και ε, η άδεια μητρότητος θα πρέπει ε, να ε, έχει πολλά προσόντα για την επίτευξη του στόχου μας δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να ασχοληθεί με το παιδί για να μπορέσει μπορέσει παιδί να αναπτυχθεί ε, φυσιολογικά και για να συμβάλλει και σε καλύτερη υγεία των, ε, ε, της μητέρας σύμφωνα με τις μελέτες του Παγκοσμίου, της Παγκοσμίου Οργανώσης Υγείας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο να επιτύχουμε μεγαλύτερη άδεια μητρότητος διότι επιπλέον όσο η γυναίκα θυλάζει η γυναίκα θα μπορεί να επωφεληθεί, θα προλάβει ορισμένες ασθένειες στο παιδί της σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ε, θα έχει και μια πιο στενή σχέση ε, με το το παιδί πράγμα το οποίο διαφυλάσσει τα δικαιώματα του παιδιού. Χρειάζεται λοιπόν να επεκταθεί η άδεια αυτή κατά δύο εβδομάδες ε, ε, που είναι ε, μία μικρή περίοδο σε σχέση με ε, τα ωφέλη για τη μητέρα και το παιδί. Εάν δεν ε, μπορέσει κανείς να βοηθήσει τα παιδιά όταν ακόμη είναι μικρά, τότε το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο αργότερα. Γι' αυτό και συνέκρινα το κόστος και τα ωφέλη σε κοινωνικό, ε, οικονομικό επίπεδο από την πλευρά του εργοδότη και από την πλευρά της εργαζόμενης. Εδώ είμαστε στην ε, Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών και Απασχόλησης. Η επίπτωση λοιπόν της ε, παράτασης της άδεια μητρότητος και βελτίωσης των όρων αποζημιώσεως θα συμβάλλουν ή στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε, μια καλύτερη, σε ένα καλύτερο συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Όσον αφορά την άδεια των ε, γονέων, ε, γονική άδεια θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό στοιχείο και θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν ευθύνες όσον αφορά τα παιδιά και ε, την περίθαλψη των παιδιών. Και οι δύο γονείς θα πρέπει να μπορούν ε, να ε, συνδυάσουν την επαγγελματική τους με την οικογενειακή τους ζωή, δηλαδή θα χρειαστεί να περιλάβουμε στην οδηγία και την άδεια πατρότητος. Θα προσπαθήσω να βρω μία καλύτερη διατύπωση με τη βοήθεια των συναδέλφων μου για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε την άδεια στην οδηγία. Θα ήθελα βέβαια να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των μελών της Επιτροπής μας, όχι μόνο επ' αυτού του θέματος, αλλά και γενικότερα. Και θα ήθελα επίσης η δικιά σας προσέγγιση να λάβει υπόψη ε, το γεγονός ότι το κόστος της άδειας ε, μητρότητος στα κράτη-μέλη μπορεί να θεωρηθεί σαν μία επένδυση και όχι σαν ένα έξοδο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρνικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι με τα μεγάλη χαρά συζητάμε αυτή την οδηγία και βεβαίως συμφωνούμε με οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την απασχόληση των εγγύων γυναικών Χωρίς όμως να επεκταθώ θα αναφερθώ στις τροπολογίες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν πρέπει η πρόθεση αυτή των εγγύων γυναικών ή των γυναίκων που θυλάζουν τις εμποδίσει να καταλάβουν μια θέση εργασίας. Μπορεί να έχουμε θαυμάσιες ιδέες, να θεωρήσουμε ότι θα βελτιωθεί η εργασία τους και στο τέλος να είναι μπούμεραν και να μην μπορέσουν οι γυναίκες αυτές κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Θα ήθελα λοιπόν το κείμενο αυτό να ασχοληθεί ουσιαστικά με τις γυναίκες γιατί ξέρω αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ε, άδεια και για τους άντρες αλλά συνήθως βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους άντρες χωρίς να τις βελτιώνουμε για τις γυναίκες και γι' αυτό επειδή καθυστερούμε πάρα πολύ θα ήθελα περισσότερο να προωθήσουμε τις γυναίκες προτού δώσουμε επιπλέον δικαιώματα στους άντρες. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες τις οποίες έχετε προτείνει, στην τροπολογία 4 σχετικά με την αποκλειστική πρόορη, ε, θυλασμό, δεν ξέρω τι εννοείται με πρόορο θυλασμό, καταλαβαίνω ότι είναι ο αποκλειστικός θυλασμός, όχι όμως ο πρόορος και ε, αυτό μέχρι δύο χρονών θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Είμαι σκεπτική διότι ε, έχουμε πολλούς γιατρούς που λένε κατά τους πρώτους μήνες, τους πρώτους τρεις μήνες τουλάχιστον, αλλά μέχρι δύο χρόνια πιστεύω ότι ε, είναι αμφισβητήσιμο. Και άντε να πάμε στους έξι μήνες. Επίσης ε, πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε ότι όλα αυτά είναι καλά μπορεί να κατά αυτόν τον τρόπο να στραφούμε κατά των γυναικών οι οποίες δεν μπορούν να θυλάσουν ε, είναι μια ε, βολή για την γυναίκα και να πούμε ότι την κάνει να αισθανθεί καλύτερα με το παιδί της χωρίς να υποχρεώσουμε τις γυναίκες όνει και καλά να θυλάζουν μέχρι δύο χρονών τα παιδιά τους. Όσον αφορά την κατάσταση στα κράτη-μέλη, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, να μην ε, αποτελέσει το μέτρο αυτό τροχοπέδι στην ε, απασχόληση και στην πρόσληψη των γυναικών και να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται στη Σκανδιναβία όπου έχουμε καλό ποσοστό γονιμότητος με μέτρα συμβιβαστικά τα οποία δεν προωθούν την παραμονή της γυναίκας ε, στο σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν ε, άλλες ρυθμίσεις ε, οι οποίες δεν πρέπει να οδηγήσουν τις γυναίκες πίσω στο να αποκλειστούν στο σπίτι. Επίσης αυτή η οδηγία προσπαθεί να βελτιώσει τους όρους εργασίας των γυναικών εργαζομένων αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι τέτοιο διότι αυτός είναι ο λόγος υπάρξεως του κειμένου αυτού. Άρα δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε και σε αυτό το σημείο λέμε ότι για τις υπόλοιπες γυναίκες οι οποίες παραμένουν ή επανέρχονται στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω τι εννοεί ε, για επάνωδο, όταν μιλάει για επάνωδο στην αγορά εργασία. Στην τροπολογία 13 λέγεται ε, να να εργάζεται κανείς όταν είναι έγκυος αλλά σαν και εκεί βοηθός domestic domestic είναι ε, ένας όρος περίεργος στη Γαλλία ίσως είναι λάθος μετάφραση αλλά ε, οι οικιακοί βοηθοί είναι αμοιβόμενες άρα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλο τον κόσμο αν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ε, έχουμε τώρα μία μία οδηγία που συζητείται στο Συμβούλιο για τις Ελεύθερες Επαγγελματίες και δεν βλέπω γιατί προσετέθη αυτό το στοιχείο. Όσον αφορά το ε, ε, ε, ε, την υγεία των εργαζομένων ε, καλύπτεται από μία άλλη οδηγία άρα δεν βλέπουμε για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η τροπολογία όταν μιλάμε επίσης για ισότητα των ανδρών και των γυναικών θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ πρόκειται για ένα κείμενο ιδίως για τις γυναίκες για να τις προστατεύσουμε και όχι για να προωθήσουμε τους άντρες όσον αφορά την ε, διάρκεια της αδείας εγώ δεν συμφωνώ να επεκταθεί η άδεια στις 20 εβδομάδες και προτείνω όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει τουλάχιστον στις 18 εβδομάδες και από εκεί ε, θα δοθεί η διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν το θέμα κατά περίπτωση. Επίσης όσον αφορά τους 27 μήνες πριν και μετά την άδεια η τροπολογία αυτή ε, αντιφάσχει με την αιτιολογία της όπου λέγεται ότι η ε, γυναίκα μπορεί να διαλέξει πόσες εβδομάδες θα λάβει πριν και μετά τον τοκετό ενώ σε ένα άλλο σημείο μιλάνε για αριθμό μηνών πριν και μετά. Ε, ας αφήσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στην μητέρα διότι υπάρχουν γυναίκες γυναίκες οι οποίες αισθάνονται πολύ καλά όταν είναι έγκυες και μπορούν ε, να εργάζονται είτε μέχρι μία εβδομάδα πριν ε, γεννήσουν ή μέχρι τον τοκετό για να έχουν περισσότερο χρόνο μετά και θα, πρέπει να τους αφήσουμε αυτή την ευχέρεια. Όσον αφορά την τροπολογία του 29, μία επέκταση αδείας ενός ε, κατά ένα μήνα ανά παιδί είναι θέμα επικουρικότητος πρέπει να παραμείνει στα κράτη μέλες. Όσον αφορά την άδεια μητρότητος, η θέση μου είναι αρνητική. Πιστεύω ότι υπάρχει μία παθολογία η οποία καλύπτεται από την εγκυμοσύνη και δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθούμε σε ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, όσον αφορά τις ε, ελεύθερες επαγγελματίες, θα πρέπει πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει μία ιδιαίτερη οδηγία για τις ελεύθερες επαγγελματίες επειδή το πρόβλημα εδώ πρέπει να παραμείνει χωριστό και να το επεξεργαστούμε ε, σε μία άλλη οδηγία όσον αφορά τις οργανώσεις και τα νομικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούν την οδηγία δεν ξέρω αν υπάρχουν οργανώσεις ε, ε, όταν ε, υπάρχουν νομικά κείμενα δεν βλέπω γιατί να προσθέσουμε εδώ την εμπλοκή των οργανώσεων. Επίσης στην τροπολογία 47 όπου λέγεται ε, ε, ότι θα πρέπει να αναφέρονται στις συλλογικές συμβάσεις και ε, τη συμβάσεις εργασίας αλλά εφόσον υπάρχει νομοθεσία δεν χρειάζεται κανείς να αναφερθεί σε άλλες παραμέτρους πρέπει να υπάρξει ούτως ή άλλως η συνθήκη εργασίας η οποία προσφέρει προσόντα και το ίδιο ισχύει και για τη συλλογική σύμβαση. Ε, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις τροπολογίες διότι θέλω επίσης να πω ότι όλα τα κράτη-μέρη δεν είναι στο, σε ίση θέση όσον αφορά τα δικαιώματα της αδείας μητρότητος. Δηλαδή ε, σε ορισμένες χώρες η άδεια μητρότητα τόσο μπορεί να θεωρηθεί σαν πλήρης χώρος απασχόλησης και να διατηρήσει η μητέρα όλα τα δικαιώματά της, η κυρία Στρό. Εστρέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συστηθώ. Είμαι αναπληρώτρια στην Επιτροπή αυτή, αλλά είμαι εισηγήτρια στην Αρμόδια Καθήλια Επιτροπή για το θέμα αυτή, Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό της αναθεώρησης αυτής τη οδηγία που είχε ήδη απασχολήσει και την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ήταν αρκετά ταραγμένη η πορεία της, γιατί ξεκίνησε με μια αναβολή της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Ε, εξακολουθώ να είμαι συγγήτρια της έκθεσης αυτής στην αρμόδια κατουσία επιτροπή και θα ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Καταρχήν, η οδηγία αυτή είναι 17 ετών είναι πια παροχημένη. Έχει φάει τα ψωμιά της. Και αν όλα πάνε καλά, η αναθεωρημένη οδηγία θα τεθεί σε ισχύ μετά την λήξη αυτής της α, κοινοβουλευτικής θητείας. Δηλαδή δεν νομοθετούμε α, για κάτι που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή αλλά νομοθετούμε για κάτι που θα τεθεί σε ισχύ τις επόμενες δεκαετίε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμόσουμε την νομοθεσία στην πραγματικότητα και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και στις ανάγκες της κοινότητα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το πεδίο εφαρμογή της οδηγία αυτής διευρύνθηκε. Ο στόχος της είναι τριπλός. Πρώτον, η προστασία της υγείας της μητέρας και η εξασφάλιση ε, της ε, ασφάλειάς της στην χώρα εργασίας, αλλά και η πρόθεση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, η διεύρυνση της νομικής βάσης, ο συνδυασμός του άρθρου 137 που αφορά την ε, υγεία με το άρθρο 141 που προωθεί την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων διευρύνει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, αυτό ο συνδυασμό των νομικών βάσεων και επιτρέπει τη συμπερίληψη και τη άδεια πατρότητα. Διευκολύνει δηλαδή το συνδυασμό τη επαγγελματική σταδιοδρομία με την οικογενειακή ζωή και για τι γυναίκε και για τους άνδρες. Επίσης, δίνει αξία και αναβαθμίζει ένα νέο μοντέλο γονιών που και οι δύο εργάζονται γιατί η αγορά εργασίας και η κοινωνία πολύ συχνά ακόμη ε, συνδέουν τη γυναίκα με τη μητέρα, κάτι που δεν συμβαίνει με τον άνδρα. Συνήθως ο άνδρας συνδέεται με την έννοια του εργαζόμενου που στηρίζει την οικογένεια με το πολιστικό επάγγελμά του και περισσότερο η κοινωνία συνδέει την ε, γυναίκα με την αναπαραγωγή παρά με την παραγωγή. Ενώ θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις δύο πτυχές. Η οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εργαζόμενες γυναίκες. Ακόμη και τις ασυνήθιστες μορφές εργασίας, τις άτυπικές. Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις της προλαλήσας σας, σε ό,τι αφορά τις οικιακές βοηθούς, πρόκειται για μια σύσταση της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας γιατί οι οικιακές βοηθοί αποκλείονται από οποιαδήποτε προστασία μητρότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες χώρες δεν εξασφαλίζουν αυτή την προστασία. Αλλά εμείς δεν νομοθετούμε για την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Νομοθετούμε για 27 χώρες μέλη. Και σήμερα η νομοθετική πραγματικότητα είναι ποικιλόμορφη. Ε, η περίοδος ε, της άδειας ε, μητρότητας κυμαίνεται από 14 σε 52 εβδομάδες στις χώρες μέλη και μερικές φορές στην άδεια αυτή μητρότητα λαμβάνεται πλήρης μισθός ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αμοιβή είναι συμβολική στη διάρκεια της άδεια μητρότητα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί η αρχή της πλήρους αμοιβή, γιατί δεν θα πρέπει η τεκνοποίηση να επιδεινώνει την οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης αμοιβή στη διάρκεια της άδεια πατρότητας ή μητρότητας και θα πρέπει τα μέτρα μας να συνάδουν με το στόχο αυτό. Φυσικά μακάρι να καταλήξουμε σε συμφωνία όσο πιο ευρία γίνεται προκειμένου να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα και στις 27 χώρες μέλη ως κοινό παρανομαστής. Γιατί υπάρχει μια ρήτρα διασφάλιση στην οδηγία αυτή που προβλέπει ότι σε περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία είναι πιο ευνοϊκή υπερισχύει η πιο ευνοϊκή νομοθεσία. Οπότε οι χώρες μέλη που έχουν ήδη μια καλή νομοθεσία, καλύτερη από αυτή που προτείνουμε εμείς, η νομοθεσία αυτή η ευνοϊκότερη υπερισχύει της κοινοτική και εξακολουθεί να ισχύει. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά είμαι και αναπληρώτρια και αυτή τη Επιτροπή και νομίζω ότι είχα δικαίωμα να σα εκφέρω τι απόψει μου και ω αναπληρώτρια εδώ, αλλά και ω συζητήτρια στην αρμόδια κατουσίαν Επιτροπή η άδεια μητρότητα θα πρέπει να συνδυαστεί με την άδεια, άδεια πατρότητα. Αλλιώ δεν προστατεύει τι γυναίκε στην αγορά εργασία. Γνωρίζουμε ότι πολλέ γυναίκε διακόπτει, διακόπτει ο πρόεδρο, γιατί έχουμε πολλού ε, ομιλητέ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Στρέλα. Καλά, θα προσπαθήσω. Θα φροντίσω να συντομεύσω. Είναι σημαντικό λοιπόν για να εξασφαλίσουμε το συνδυασμό της επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή να συμπεριλάβουμε στην οδηγία και την άδεια πατρότητας που δεν έχει καμία σχέση με τη γονική άδεια γιατί η γονική άδεια είναι αντικείμενο άλλης οδηγίας. που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και περιμένουμε σύντομα πρόοδο και στο θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια καινοτόμα πρόταση, απέτηση των καιρών, να συμπεριληφθεί και η άδεια πατρότητα στο πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ευχαριστώ. θα Νομίζω ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε όλοι. Γιατί έχουμε 8 ομιλητέ ακόμα. Και θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει και η ομιλήτρια, η κυρία Χάρ. Και μετά η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και την εισηγήτρια ευχαριστώ. Δεν άκουσα όλη τη συζήτηση αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση για μένα. Η ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απλώς ένα συμβιβασμός διότι τα κράτη-μέλη θα δουν αν θέλουν να υπερβούν την οδηγία ή όχι. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο για την προστασία της υγείας και ιδίως για τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν αμέσως στην εργασία να έχουν χρόνο να κατατίσουν μία στενή σχέση με το παιδί και ε, να προχωρήσουν. Επίσης μετά από 20 εβδομάδες νομίζω ότι στην ε, περίοδο οικονομικής κρίσης θα είναι δύσκολη η κατάσταση και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόδιο διότι ε, οι γυναίκες ε, ίσως δεν θα μπορούν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά ή δεν θα βρίσκουν θέση. Ε, πρέπει λοιπόν να ζυγίσουμε στην οδηγία αυτή τα δικαιώματα των εγγύων και νέων μητρών, μητέρων χωρίς όμως να επιδεινώσουμε την θέση εργασίας. Εδώ όντως η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι η οι μέρες ασθενείας για εγκυμοσύνη δεν θα συνυπολογίζονται αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στις, με τις 18 εβδομάδες για να είναι προστατευμένος και ο εργαζόμενος. Επίσης νομίζω ότι καλό είναι να μπορεί η μητέρα να διαλέξει πότε θέλει να πάρει την άδεια μητρότητός της και ε, χρόνος αδείας ε, για τους γονείς, γονική άδεια δηλαδή που υπάρχει σε ορισμένα κράτη θα πρέπει να γενικευθεί, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Ε, είναι βασική η άδεια μητρότητος αλλά πρέπει απλώς να βελτιώσουμε την σχέση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής χωρίς όμως να αποτελέσει αυτό φραγμό στην απασχόληση των γυναικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό συζητήθηκε ε, επαρκώς και γι' αυτό θα είμαι σύντομη. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η προστασία και η σχέση με την προστασία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε κάτι που ήδη ελέγχθη. Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια χωρίς ε, να δημιουργούμε προβλήματα στην απασχόληση των νέων γυναικών. Γι' αυτό και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό είναι το ένα σχόλιο μου. Το άλλο σχόλιο αναφέρεται στην γονική άδεια και το εάν θα πρέπει στην οδηγία αυτή να συμπεριληφθεί η γονική άδεια. Διότι όντως υπάρχει μια τέτοια επιθυμία όταν μιλάμε για ισότητα ευκαιριών. Δηλαδή θα είναι ένα θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αλλά σε αυτήν την οδηγία μας απασχολεί η υγεία και η ασφάλεια. Μέχρι όταν αρχίσουν να γεννάνε οι άντρες δεν μπορούν να προστατεύονται στον ίδιο βαθμό με τις γυναίκες άρα ε, πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε και την ισότητα των ευκαιριών διότι εδώ η βιολογία μας ε, θέτει τα όρια Όσον αφορά την ε, γονική άδεια, ε, και εδώ αναφέρουμε στη γονική άδεια, όχι στην ε, άδεια μητρότητος, υπάρχει όμως μια χωριστή οδηγία κατόπιν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και το Συμβούλιο έχει αποφανθεί. Επ' αυτού το Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να σημειώσουμε ότι επετεύχθη συμφωνία δηλαδή το θέμα της άδειας πατρότητος δεν πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταρτίζει ε, καταρτίζει νομοθετήματα για την ε, πατρική άδεια, άρα δεν είναι εδώ το κατάλληλο σημείο να συζητηθεί. Όσον αφορά την επιστροφή στην εργασία, έχω ακόμη ένα σχόλιο σχετικά με ε, τις τροπολογίες 31 και 33 και ιδίως την 33. Η ύφεση είναι μία μάλλον η κατάθλιψη με συγχωρείτε είναι μια ιατρική γνωμάτευση και άρα δεν μπορούμε να το περιλάβουμε χωρίς να περιληφθεί ε, στο ιατρικό θέμα στην ε, ε, στην οδηγία. Η επόμενη ομιλήτρια θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, θα μιλήσω όμως δανέζικα θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι ε, η ισχυώδη συγγήτρια των Πρασίνων αλλά την αντικαθιστώ. Είναι βασικό, βασική αυτή η οδηγία για τις γυναίκες, για την υγεία τους και για τις δραστηριότητές τους στην αγορά εργασίας Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μία Ευρώπη με μεγαλύτερη γεννητικότητα θα πρέπει να επιτρέψουμε στις γυναίκες να κάνουν περισσότερα παιδιά και να συνδυάσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Μιλάμε πολύ για το κόστος της δημογραφικής εξ, ε, της εξελίξεως αλλά καταρχήν θα πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να έχουν παιδιά. Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε στη διάρκεια της αδείας μητρότητος. Εδώ η συγγήτρια μιλά για 20 εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 18. Στη Δανία όμως μπορείτε να έχετε ένα ολόκληρο χρόνο ε, της ε, αδείας μεταξύ της μητρικής και πατρικής αδείας και η κυρία Εστέλα είπε πολύ σωστά τι έχει κάνει αλλά εδώ δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι άντρες μπορούν να πάρουν άδεια πατρότητος στην Δανία αλλά δεν τη χρησιμοποιούν. Υπάρχει όμως υποχρεωτική άδεια τριών μηνών και η άντρες υποχρεώνονται να την ε, λαμβάνουν. Εάν ε, ε, μείνουμε στις 18 ευρωμάδε για την άδεια μητρότητος για τις μητέρες, οι άλλες δύο ως τις 20 θα μπορεί να είναι άδεια πατρότητος, για τους άντρες δηλαδή. Επίσης ένα μέρος της αδείας μπορεί να ληφθεί πριν τον τοκετό. Εδώ όμως πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθεί κανείς στην περίοδο μετά το δοκετό για διάφορους λόγους γιατί δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η κυρία Στέλ και μετά ο Τόμας Μάν. Συμφωνώ απόλυτα με την προλαλή σας, την Έμιλη, εκ μέρους των Πρασίνων. Υπάρχει ένα τμήμα της προστασίας των γυναικών σε σχέση με την υγεία και το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την έγκυο, τη μέλουσα μητέρα, αλλά να προστατεύσουμε και το παιδί που θα γεννηθεί. Στις εργασιακές συνθήκες σήμερα, πολλές φορές η ε, ατμόσφαιρα της επιχειρήσης, ο αέρας της επιχειρήσης είναι γεμάτος ε, ε, χημικές ουσίες που διαταράσσουν και την, τον ενδοκρινολογικό σύστημα. Και πολλές φορές ε, όταν σε μια τέτοια ατμόσφαιρα στάνει μια έγκυος αναπνέει αυτές τις χημικές ουσίες ε, που διαταράσσουν ε, την ορμονική ισορροπία της. Αυτό το θέμα λοιπόν του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας δεν αναφέρεται σε σχέση με την υγεία των έγκυων. Οι γυναίκες που εργάζονται στα στεγνοκαθαριστήρια, αναπνέουν επικίνδυνες χημικές ουσίες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πώς λοιπόν θα προλάβουμε τέτοιου είδους θέματα. Προτιμώ να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης στις επιχειρήσεις για τις εγγύους. Και μάλιστα βρήκαμε κάποιες τροπολογίες που προλαμβάνουν αυτό το θέμα, ώστε όλες αυτές οι χημικές ουσίες και τα αέρια, που είναι και καρκινογόνες, να περιορίζονται στον αριθμό για να προστατεύονται οι έγκυες γυναίκες. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορούμε, πώς μπορούμε να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τις έγκυες γυναίκες από, σε αυτό το επιβλαβές περιβάλλον. Uh, thank Σας ευχαριστώ. Τόμας Μάνο. Και μετά κύριε Φιρέιδο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου Έχετε δίκιο ότι εσείς ε, κατέχετε το θέμα, αλλά στα θέματα ανατροφής ε, παιδιών παίζουν φυσικά και ένα μικρό ταπεινό ρόλο και οι άντρες. Και να πω ότι ήμουνα και εγώ επί 10 έτη μέλος της ε, Επιτροπής για την Ισότητα των φίλων και αισθανόμουν πάντα μια χαρά. Νομίζω ότι επί της αρχής συμφωνούμε, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και φυσικά και το κόστος παίζει ρόλο του. Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αρχή της ε, σύνδεσης και της συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και οικογένειας, προκειμένου οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα και να κάνουν παιδιά, αλλά και να έχουν ε, μια σωστή σταδιοδρομία και να υπάρχουν και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Και συμφωνώ, όπως είπε και η κυρία Μπάουερ, ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα ε, με μία οδηγία. Το θέμα, για παράδειγμα, με την οδηγία για τις αντιδιακοπών ε, είναι άλλο θέμα, να μην τα μπλέκουμε. Θεωρώ ότι σωστά λέτε στην τροπολογία 7 ότι και σε εμά στη Γερμανία θα πρέπει οι 14 εβδομάδες που προβλέπονται για άδεια μητρότητας, 6 εβδομάδες πριν από την ε, γέννα και 8 εβδομάδες μετά τη γέννα, ε, προτείνετε όμως τώρα 20 εβδομάδε και λέτε ότι είναι πιο σημαντική η επένδυση παρά το να μιλήσουμε τα οικονομικά μα. Και αυτό το είπαν και κάποιε άλλε ομιλήτριες, ότι αυτό δεν μπορεί να καταστεί εμπόδιο. Γιατί υπολογίσαμε τα εξή. Αν γίνει μια αλλαγή στη Γερμανία από 14 σε 20 εβδομάδε στη Γερμανία, μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προστιθούν. Πώς θα το περάσουμε αυτό πώ θα συνδυαστεί αυτό με τα συμφέροντα των κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο το χρειαζόμαστε, γιατί νομίζω ότι σε κάποιες λεπτομέρειες απέχουν αρκετά οι θέσει μας. Θα χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο, αλλά το προωθεί πάρα πολύ γρήγορα η Επιτροπή Γυναικών και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε. Τελευταία παρατηρήση. Λέμε ότι θέλουμε ένα μέσο κατά της κρίσης, σημαντικό και αυτό. Αλλά να δούμε ότι υπάρχει και μία φάση, αν θέλετε, μεταβατική, η οποία θα είναι αρκετά ικανή για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε το νέο μέτρο αυτό. Γιατί αυτή η σαφής αλλαγή από 14 σε 20 εβδομάδες νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και η Κομισιόν προτείνει 18 εβδομάδες. Είναι, πιο, είναι λιγότερο έντονη η διαφορά. Νομίζω ότι με μια κοινή συζήτηση θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Φιγκρίδο. Σας ευχαριστώ. Δύο σύντομα σχόλια, γιατί έγινε εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό. Τα δύο ουσιαστικά ζητήματα είναι τα εξής. Θέλουμε να αυξήσουμε ή όχι τον αριθμό των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το θέλουμε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη μητρότητα, τη μητρότητα και την πατρότητα. Θα πρέπει να συνδυάσουμε όχι μόνο την αύξηση της γεννητικότητας, ε, αλλά και την ανάγκη εξασφάλισης ισότητας δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών φυσικά θα πρέπει να είναι ευθύνη της μητέρας και του πατέρα. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Γι' αυτό και το να περιλάβουμε την άδεια πατρότητα στην οδηγία είναι πολύ λογικό. Αν θέλουμε να προσπίσουμε και την ισότητα των δύο φύλων, αλλά και τα δικαιώματα του παιδιού. Γιατί έτσι θα απολαύσει την παρουσία και του, των δύο γονιών του, ήδη από την ε, μικρή του ηλικία, από την τρυφερή ηλικία. Επίσης υπάρχουν εδώ κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Και εκ μέρους της ΓΚΟΕ θα υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια εγγύηση για την προθεσμία για την απόλυση των εγγύων γυναικών ή των γυναικών που έχουν γεννήσει. Θα πρέπει να αποκλείεται η απόλυση γυναικών που έχουν γεννήσει τουλάχιστον για ένα χρόνο. Επίσης θα πρέπει οι άδειε μητρότητας και πατρότητας να είναι άδειε θα πρεπει οι αδειε και πατροτες να ειναι πλήρους αμοιβής παρόλο που υπάρχει μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, τουλάχιστον θα πρέπει στην διάρκεια της άδεια οι δύο γονείς να λαμβάνουν το μισθό τους ακέραιο. Και τέλος, θα να πω ότι η οδηγία αυτή, όπως ξέρουμε, ισχύει εδώ και 20 χρόνια. Είναι οδηγία το 85. Προτείνουμε τώρα την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας ε, για το μέλλον. Δεν θα ισχύσει μόνο στο παρόν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και διορατικοί. Γιατί η κρίση καταπολεμάται και με τη βελτίωση της κοινωνικής στήριξης και προστασίας. Αυτό θα είναι μια επένδυση ε, στο μέλλον και όχι μια δαπάνη και ένα κοινωνικό άχθος. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να ξεφύγουμε από την κρίση και η οδηγία αυτή θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά τα οποία πολύ σωστά είπαν ε, ο Πασκάλ Γιονί η Έντιτ Μπάουερ και ο Τόμας Μαν, αλλά θα ήθελα να τονίσω τρία θέματα. Καταρχήν, το κείμενο αυτό είναι καλό για τη βελτίωση της, ε, ασφάλεια ασφάλειας και της ε, υγείας των εγγύων γυναικών, των λεχόνων και των γυναικών που θυλάζουν. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα χωρίς να αναμειγνύουμε και άλλα γιατί αντελήφθηκα ότι σιγά σιγά παρεκκλίνουμε προς άλλα θέματα δεν αναφέρουμε στην άδεια πατρότητος αλλά όσον αφορά την, ε, την ε, ανατροφή των παιδιών θα μπορούσε κανείς να προσθέσει πολλά άλλα πράγματα οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ε, το αρχικό στόχο μας. Δεύτερον, ε, είμαι υπέρ και το λέω εδώ και πολύ καιρό της, του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αλλά εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γυναίκες, ε, οι έγκυοι ή οι φυλάζουσες ε, που επιστρέφουν στην δουλειά τους πρέπει πρέπει να μπορούν να βρουν δομές οι οποίες να τους επιτρέψουν να συνδυάσουν ε, το θυλασμό, την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Χρειάζονται λοιπόν υποδομές για να στηριχτούν οι γυναίκες αυτές κατά την ε, εργασία τους. Επίσης, η άδεια μητρότητος. Βεβαίως θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την άδεια μητρότητος και θα είχαμε όλο και περισσότερο ε, γυναίκες οι οποίες θα ήθελαν να κάνουν παιδιά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι. Ε, η παράταση της άδειας μητρότητος, αν γίνει αλόγιστα, θα είναι εις βάρος των γυναικών για την επιστροφή τους στη δουλειά. Η επαγγελματική ζωή αλλάζει και εάν εάν επεκτείνουμε την άδεια μητρότητος δυναμητίζουμε την επιστροφή στην εργασία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με την διάρκεια της αδείας μητρότητος κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να επεξέλθουμε τις κρίσεις. Ευχαριστώ. Και τελικά η κυρία Σάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποδείχτηκε ότι η εθνική νομοθεσία σε πολλές χώρες για τις διατάξεις, ε, μάλλον ξεπερνάει τις διατάξεις της οδηγίας αυτής και όπως είπε και η κυρία Μπάουερ, πέφτει για ένα ελάχιστο όριο, μια ελάχιστη οδηγία. και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο τροπολογίε όπου υπάρχουν πραγματικά νομικά προβλήματα και σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα κάποιων χωρών. Το πρώτο από αυτά τα σημεία σχετίζεται με την τροπολογία υπερθυμών 41 που αναφέρεται. ότι ένας γονιός ή ένας από τους δύο συζύγους μάλλον ο σύζυγος της εν λόγω μητέρας μπορεί να ζητήσει άδεια πατρότητος. Αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό γιατί δεν μπορούμε να περιορίσουμε, να μεταβιβάσουμε το δικαίωμα αυτό της γυναίκας ε, σε ένα άλλο άτομο όσο και έντονη αυτή είναι η επιθυμία. Για παράδειγμα στη Φιλανδία δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί το δικαίωμα αυτό σε άλλο άτομο. Πρόκειται για θέμα συνταγματικό το οποίο τίθεται. Και θα τίθεται φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Και στην τροπολογία υπαριθμών 40 που αναφέρεται. Ότι ρυθμίζεται επακριβώς η αμοιβή που χορηγείται ότι δεν πρέπει να, υπερβαίνει, δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο του 85%. σε πολλές χώρες αυτό δεν είναι θέμα μόνο του, εργα... εργοδότη. Είναι και θέμα κοινωνικής ασφάλισης. Άρα θα πρέπει να λεφθούν υπόψη και οι διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των ε, κρατών μελών και σε κάποιες χώρες είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι εδώ και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Αυτά τα δύο στοιχεία, αυτές οι δύο τροπολογίες υπαριθμών 40 και 41 είναι προβληματικές θεωρούμε, γιατί τίθεται θέμα αρμοδιότητας. Και αυτό αντίκειται και στην εθνική νομοθεσία μάλιστα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η εισηγητρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στη συζήτηση αυτή. Να απαντήσω το Σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, ε, μητέρων στον χώρο εργασίας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, όλα αυτά σχετίζονται με τις συστάσεις της Διεθνούς ε, οργάνωσης, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. το γεγονός ότι στην οδηγία αυτή υπάγονται όλες οι εργαζόμενες ανεξάρτητα από την σύμβαση εργασίας τους Κοιτάξτε, αυτό το θέμα που τίθεται για τις ε, οικιακές βοηθούς αυτή τη λέξη, αυτόν τον όρο χρησιμοποιούμε για τις γυναίκες που απασχολούνται στο ιστορικό ενός Και τον όρο αυτό χρησιμοποίησαμε και στην προηγούμενη θητεία. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτός ο όρος να μεταφραστεί να μεταφερθεί και στα γαλλικά. Και σε αυτόν τον όρο, ε, σε αυτόν τον όρο, στον ορισμό καταλέγονται και όλες οι συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις συστάσεις της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του ILO. Στη συνέχεια, θέλουμε να πετύχουμε κάποιες βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την οδηγία αυτή. Και αυτό είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά σε συνάρτηση και με την τρέχουσα κρίση. Να τονίσω λοιπόν το εξή. Να θεωρήσουμε ότι πρόκειται όχι για κρατική δαπάνη, αλλά για επένδυση. Γι' αυτό λοιπόν να παρακαλέσω τους συνοδέλφους το εξή. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να βρούμε τις καλύτερες λύσεις, την καλύτερη δυνατή λύση για να εξέλθουμε τις κρίσεις. Και είμαι αισιόδοξη, είμαι βέβαιη ότι πρόκειται να την ξεπεράσουμε την κρίση αυτή. Θα πρέπει να δούμε προκειμένου με την ε, οδηγία αυτή σε επίπεδο κρατών μελών να ακολουθήσουν συγκεκριμένα μέτρα σε διάστημα 2 ή 3 ετών. Θεωρώ ότι μόνο τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ξεπεράσει την σημερινή κρίση. Μακροπρόθεσμα μιλάω πάντα. Τώρα, για τις μεμονωμένες τροπολογίες και τα σχόλια που έγιναν. Σίγουρα θα τα συζητήσουμε αυτά με τους συναδέλφους, θα ανταλλάξουμε και email για να εξηγήσουμε ο ένας τον άλλον πιο συγκεκριμένα τις ε, προτάσεις τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και υπολογίζω στη συνεργασία σας. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα καταλήξουμε σε συνένεση. Γιατί σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την οδηγία αυτή προκειμένου να καταστεί ένα πραγματικό μέσο το οποίο θα συμβάλλει στην ε, συμφιλίωση αυτή, αν θέλετε, μεταξύ ε, εργασίας και οικογένειας, μεταξύ της ισότητας μεταξύ των φίλων. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική αρχή για την δημοκρατία, γιατί η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν λειτουργεί και η δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν και ζητώ τη συνεργασία σας και είμαι βέβαιη ότι από κοινού θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτές τις ε, βελτιώσεις που επιζητούμε και είμαι βέβαιη ότι ως Επιτροπή θα συνεργαστούμε άριστα με την Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων. Είμαι και αναπληρώτρια στην Επιτροπή αυτή και θεωρώ ότι από κοινού όντως θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις, τις καλύτερες διατυπώσεις για την προστασία των γυναικών στον χώρο εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λήγει στις 12 Νοεμβρίου το μεσημέρι. 12 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και ολοκληρώσαμε την ημερήσια μας διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει την 3η 1η Δεκεμβρίου στις 3 και την 4η 2 Δεκεμβρίου